Παρακαλώ καθίστε συνάδελφοι, θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη και μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν όπως προβλέπετε το πρόγραμμα. Πριν ξεκινήσουμε την ακρόασή μα, θα ήθελα να κάνω ορισμένες ανακοινώσεις. Καταρχάς, ο κύριος Κασουλίδης ορίστηκε ως μόνιμος εισήγητης για τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Ε, ό,τι καλύτερο κύριε Κασουλίδη. Τώρα, η... θα ήθελα να σας ενημερώσω επίσης ότι σχετικά με την απόφαση που πήρε το Προεδρείο για την ε, κατάθεση συστάσεων προς το Συμβούλιο γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ουκρανία και Γεωργία. Πρόκειται για συστάσεις οι οποίες αφορούν μία πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε συνεκτική με τις αρχές μας απέναντι σε ολοκληρωτικά καθεστώτα όπως ακριβώς το φροντίζει αυτό ο κ. Βότσον. υπήρξαν ε, για τον καθορισμό των ε, καταλόγων ψηφοφοριών υπήρξαν ε, κάποια προβλήματα πρακτικά. Θα πρέπει να κατατεθούν οι προτάσεις 24 ώρες πριν από την ψηφοφορία. δεν αποκλείεται η δυνατότητα κατάθεσης προφορικών τροπολογιών βέβαια αλλά είπαμε ότι για να αποφύγουμε τα προβλήματα που έχουν ήδη ξεκινήσει να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις. Δεν σας καθυστερήσω άλλο, περνάμε τώρα στο βασικό θέμα. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρη η παρουσία εδώ των συνομιλητών μας. Σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση με την οποία ξεκινάμε τη συζήτηση του θέματος για την κατάσταση στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Η ακρόαση αυτή έχει σαν στόχο να εμβαθύνει τις γνώσεις τις οποίες έχουμε σαν κοινοβουλευτική γύρω από το θέμα αυτό και να επιτρέψει να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση γύρω από την έκθεση Κυριλόφ για την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον Νότιο Κάφκασο. Di valutazione di discussione molto interessante, recentemente Πρόσφατα ψηφίστηκε, πέρασε και το ψήφασμα για την ανατολική διάσταση της ε, πολιτικής γειτονίας. Υπεύθυνο είναι ο κύριος Σίβιετς. Qualificati che sono ai vari livelli coinvolti nel negoziato per la soluzione del conflitto. Λοιπόν, Έχουμε μαζί μας τον κύριο πρέσβη Ρόμπερτ Μπρέτκι, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος από τις Ηνωμένε Πολιτείες της ομάδας του Μίνσκ. Έχουμε τον πρέσβη Φασιέ, επίσης Γάλλος συμπρόεδρο, τον πρέσβη Άντρεϊ Κάρπισκ, προσωπικό αντιπρόσωπο της ε, Προεδρίας του ΟΑΣΕ, και τον Πίτερ Σένμπι, τέος ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ανατολικό Κάυκασο. Συγγνώμη, τον Νότιο Κάυκασο. Δεν έχουμε μαζί μας τον Ρώσο συμπρόεδρο της ομάδας του Μίνσκ, τον κύριο Ποπόφ. Ο κύριος Ποπόφ δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας γιατί είχε ε, ταυτόχρονες ε, ανηλυμένες υποχρεώσεις. Έχουμε επίσης ε, και τον κύριο Μύρος Λαβλάιστατ θα ήθελα να τον καλέσω και αυτόν να σχολιάσει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις οι οποίες διεξάγονται. Θα συνεχίσουμε λοιπόν δίνοντας το λόγο στον πρέσβη Ρέτκε για πέντε λεπτά ίσως ίσως και λίγο περισσότερο αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να προσπαθήσουμε να μην καθυστερήσουμε πολύ και να σας δώσουμε τη δυνατότητα να απαντήσετε και στις ερωτήσεις οι οποίες θα σας τεθούν. Λοιπόν, πέντε λεπτά εάν είναι δυνατόν, αλλιώς θα δούμε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μας είχαν πει δέκα λεπτά, οπότε θα προσπαθήσω να τα συρρυκνώσω σε πέντε λεπτά. Να πω εξ αρχής ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι ανάμεσά σας σήμερα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση την οποία έλαβα από σας και την Επιτροπή σας την οποία συνάντησε η Υπουργός Εξωτερικός Κλίντον πέρυσι. Ε, συναντήθηκε και με την Επιτροπή σας και με τον Πρόεδρο Μπούζεκ φυσικά. Πιστεύουμε στις Ηνωμένε Πολιτείε ότι πρέπει να ενισχυθεί κάθε μορφή συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όχι μόνο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά αναφερθήκαμε ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικά. Η παρουσία μου εδώ αποδεικνύει ακριβώς το πνεύμα αυτής της ε, προσπάθειας. Η Υπουργό Εξωτερικών ε, συναντήθηκε και με τη Λέιδη Άστον σχετικά με την ε, εταιρική σχέση ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ ΕΕ είναι εταίροι που συνεργάζονται σε όλα τα θέματα, περιφερειακά και παγκόσμια, σε όλα. Και δεν είναι εξαίρεση φυσικά τον Αγκόρνο Κάραμπα, εμείς συνεργαζόμαστε με μια χώρα αντιπρόεδρο της ομάδας του Μίνσκ, τη Γαλλία. Συνεργαζόμαστε με τη Λιθουανία που αυτή τη στιγμή προεδρεύει στον ΟΑΣΕ. Συνεργαζόμεθα επίσης και με τους συναδέλφους στην Υπηρεσία Εξωτερικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την Γραμματεία της ε, γενικότερα πολιτικής ε, των μέσων ε, των πολιτικών που έχει θέσει στη διάθεση της περιοχής και της προσανατολάς των Ευρωπαϊκών Συνόρων Περιοχής η Ευρωπαϊκή Ένωση. πέρα από αυτά θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα σημεία. Πρώτον, μια πρώτη ενημέρωση για το καθεστώς των επαφών. Δεύτερον, να αναφερθώ στις θέσεις ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και την εμπλοκή τους στις προσπάθειες ειρήνευσης του Ναγκόνο Καραμπά. Και τρίτον, λόγω των ενδιαφερόντων σας, να αναφερθώ στον ρόλο των πιθανό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Για να ξεκινήσω με, τις, ε, με το παρόν καθεστώς των διαπραγματεύσεων. Όλοι είδατε νομίζω την δήλωση της Προεδρίας δηλαδή του Προέδρου Σαρκοζή, Ομπάμα και Μετβέντεφ που βγήκε στο Ντοβίλ. Στον Ντοβίλ και οι τρεις πρόεδροι ζήτησαν από όλες τις χώρες να κάνουν σημαντικά βήματα για την ειρήνη στον Ακόρνο Κάραμπα. Ζήτησαν να καταλήξουμε στις βασικές αρχές της συνεργασίας μας για το θέμα αυτό στην επόμενη, επόμενη συνάντηση. Ποιες είναι οι βασικές αρχές. Είναι κείμενο πλαίσιο, ένα έγγραφο πλαίσιο, το οποίο παρέχει λεπτομερείς οδηγίες προς τους υπουργούς και των δύο πλευρών και που περιλαμβάνουν τα βασικά χαρακτηριστικά ε, της ε, ε, τελικής λύσης. Δεν είναι η τελική, αν θέλετε, αποφασιστική λύση, αλλά είναι οι κατευθυντήριες γραμμές γύρω από το πώς θα πρέπει να προσωμιάζει αυτή η λύση. Έχω λεπτομέρειες εδώ, δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά παρόλα αυτά α, ασχολούμεθα αρκετό καιρό. Εδώ ο παρακαθήμενος πρόεδρος γνωρίζει το θέμα γιατί ασχολείται περισσότερα χρόνια από μένα. Νομίζω ότι επί τη βάση αυτών των αρχών θεωρούμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια ισόρροπη και δίκαιη λύση και θα θέλαμε οι εμπλεκόμενοι να δεχτούν τις προτάσεις αυτές. Δεν θα περάσω τώρα σε επίπεδο λεπτομέρειες, δεν είναι ο σωστός χώρος για κάτι τέτοιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς βασίζουμε σε έξι στοιχεία τα, την πολιτική που θα θέλαμε να ακολουθήσουμε και που περιλαμβάνονται και στη δήλωση των Προέδρων της Δοβίλ. Καταρχάς, την επόμενη συνάντηση κορυφής η οποία θα φιλοξενηθεί και θα οργανωθεί από τον πρόεδρο Μετβέντεφ. Εδώ χαιρετίζουμε τον ρόλο τον οποίο έχει παίξει ο πρόεδρος Μετβέντεφ και ο υπουργός Λαυρόφ. Έχουν επενδύσει ιδιαίτερο χρόνο σε μια δύσκολη κατά τα άλλα διαδικασία. Οι ε, Ηνωμένε Πολιτείε και από την πλευρά τους βέβαια εμπλέκονται σαφώς στην περίπτωση αυτή. Ε, συνάντησε ο πρόεδρος Ομπάμα πέρυσι και τον πρόεδρο Σαρκισάν στην Ουάσιγκτον και τον πρόεδρο Αλίεφ στη Νέα Υόρκη Υπήρξε επίσης και η πρώτη επίσκεψη της κυρίας Κλίντον στο Γερεβάν και στο Μπακού πέρυσι μετά από τις επισκέψεις που είχε κάνει ο Μπέικερ εδώ και αρκετά χρόνια. Τον Μάρτιο ο πρόεδρος, η κυρία Κλίντον συνάντησε επίσης και τον Σαρκισιάν και τον Μοχαμέντοφ ε, συνάντησε τους ε, δύο υπουργούς της Αρμενίας και της ε, άλλης εμπλεκόμενης χώρας στη Ουάσιγκτον. Ο υφυπουργό Εξωτερικών, υπεύθυνο για τα ευρωπαϊκά θέματα, επισκέφθηκε επίσης επανειλημμένα και το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ και στις δικές μας προσπάθειες εγώ διέσχισα τον Ατλαντικό από τότε που ξεκίνησα την προσπάθεια αυτή το Σεπτέμβριο του 2009 32 φορές για να συναντηθώ με τους εκπροσώπους των δύο εμπλεκομένων χωρών, με ευρωπαϊκές αρχές και με την ηγεσία του ΟΑΣΕ. Συνεπώς λοιπόν οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει μια ειρηνική δίκαιη λύση στην περίπτωση του Ναγκόρνο Κάραμπα. Να τελειώσω αναφερόμενος στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αρχή των παρατηρήσεων μου αναφέρθηκα σε ορισμένα θέματα τα οποία ήδη ε, σημειώνουν και αποδεικνύουν την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια δεν είναι δική μου δουλειά να πω σε εσά τι θα πρέπει να κάνετε. Εγώ είμαι Αμερικανός και η απόφαση αυτή είναι δική σας, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω δύο πολύ σύντομα σχόλια. Πρώτον, θεωρώ ότι ο υπάρχον μηχανισμός της ε, προσπάθειας αυτής των τριών συμπροέδρων της ομάδας του Μίνσκ είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τουλάχιστον φάση της διαδικασίας δεν είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει άμεσα βέβαια στην επίλυση του προβλήματος αλλά παρόλα αυτά προωθεί την υπόθεση και νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται και οι δύο πλευρές και αποτρέψαμε να υπάρξει αδίποτε πολεμική σύραξη στην περιοχή. Αυτό θεωρώ ότι είναι θα έλεγα κάτι το οποίο πετύχαμε σαν ομάδα του Μίνσκ. Θυμηθείτε ε, τι έχει γίνει στο παρελθόν. Η ομάδα του Μίνσκ είναι μια ευέλικτη ομάδα, επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις εξελίξεις της περιοχής, μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε το απόρριτο των διαπραγματεύσεων, το οποίο απαιτούν και οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές. Συνεπώς, εμένουν σε αυτό. Λοιπόν, είναι μια καλή διαδικασία και νομίζω ότι απέδειξε ότι είναι και μια αποτελεσματική διαδικασία. Καθώς περνάμε από αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων στην πλήρη εφαρμογή των προτάσεων αυτών, καθώς θα περάσουμε εννοώ, θα υπάρξει η δυνατότητα για όλες τις χώρες να συνεισφέρουν ακόμα περισσότερο στην ειρηνευτική διαδικασία και εδώ φυσικά ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε τις ικανότητές της σε πάρα πολλούς τομείς, στο λεγόμενο soft power. Από την άλλη πάλι δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε το ότι όσο προχωράμε στη φάση εφαρμογής θα υπάρξουν πολλές δυσκολίες και προσπάθειες που θα πρέπει να γίνουν, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και στο τέλος της διαδικασίας υπάρχει βέβαια και το θέμα της επιστροφής των προσφύγων και της ανοικοδόμησης των περιοχών. Συνεπώς όλα αυτά είναι θέματα στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Όσο προχωράει λοιπόν αυτή η διαδικασία και στο άμεσο μέλλον ελπίζω ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι και όλο και με μεγαλύτερος. Λοιπόν αυτά ήταν τα βασικά που είχα να σας πω και θα είμαι στη διάθεσή σας εκ των υστέρων να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη Μπρέτκε. Θα δώσω το λόγο στον πρέσβη Μπερνάρ Φασιέ, Γάλλο συμπρόεδρος της ομάδας του Μίνσκ. Και εσείς παρακαλώ να μείνετε στα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι η ομάδα συμπροεδρίας του Μίνσκ δεν απαρτίζεται μόνο από τρεις χώρες, Ηνωμένε Πολιτείες, Ρωσία και Γαλλία, αλλά είναι μια ενωμένη ομάδα και πολύ ενωμένη στο επίπεδο των διαμεσολαβητών, στο επίπεδο των υπουργών. Αρχικά παρουσιάσαμε τις λεγόμενες αρχές της Μαδρίτης σε πολιτικό επίπεδο με την τρόικα των τριών υπουργών και επίσης στο επίπεδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων την λεγόμενη δήλωση του Ντοβίλ, η οποία ήταν η τρίτη δήλωση μεταξύ Ομπάμα, Μετβέτεφ και Νικολά Σαρκοζή. Και στο πλαίσιο της Ενωμένης ε, Τρόικα και ξεκινώντας μία εργασία που διαρκεί εδώ και 6,5 χρόνια, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συγχωρέσετε την απουσία του Εγκόν Βαλεντίνοβιτς Ποπόφ, του Ρώσου φίλου μας, ο οποίος έχει ενημέρωση υποχρεώσεις για την ε, προετοιμασία της επόμενης ε, σημαντικής στιγμής των διαπραγματεύσεων της προσεχής εβδομάδες ε, που θα γίνει σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Η πρόθεσή μου είναι να δείξω τρία σημεία. Πρώτον, ο Μπομπ Μπράτκι σας είπε κάποια πράγματα για το τρέχον επίπεδο των διαπραγματεύσεων. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε το τι έγινε πριν γιατί η κατάσταση που έχει σήμερα είναι η έκβαση μιας, ιστορικής, μιας εξέλιξης. Δεύτερον, θα αναπτύξω κάποιους λόγους που εξηγούν το πώς η παρούσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων λειτουργεί αποτελεσματικά και τρίτον θα αναπτύξω ορισμένες παρατηρήσεις σε σχέση με, την, με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν, όσον αφορά τις διαπραγματεύσει, θα πρέπει να γνωρίζετε το λίγο πολύ οι διαπραγματεύσεις αυτές ε, αποτελούν το τρίτο μεγάλο κύκλο διαπραγματεύσεων. Μετά την εκεχηρία είχαμε τον πρώτο κύκλο, τον πρώτο γύρο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι διαμεσολαβητές της εποχής εκείνης προσπάθησαν να επανεντάξουν τον Αγκόρνο Καρεμπάχ στη διοικητική δομή του, του Αζερβαϊτζάν. Αλλά η προσπάθεια αυτή απέτυχε γιατί θεωρήθηκε σαν ένα δυνατό κάζους μπέλι ε, για την Αρμενία. Στη δεύτερη φάση, στο δεύτερο γύρο, το τέλος της δεκαετίας του 1990, ε, αρχές του 2000, οι διαμεσολαβητές προσπάθησαν να φανταστούν μια λύση η οποία θα καταστήσει δυνατή την επισημοποίηση της ε, απόσχησης του Αζερβαϊτζάν με έναν αποδεκτό τρόπο από τον Μπακού. Και αυτό απέτυχε και θεωρήθηκε κάζους μπέλη από τον Μπακού. Ο λόγος για τον οποίο ο τρίτο, στον τρίτο γύρο, τον παρόντα γύρο, εμείς ε, προσπαθούμε με τους ε, προκατόχους, το Ρώσο και το Αμερικανό συνάδελφο, να μην ε, κάνουμε μια οριστική προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης, αλλά καταρχήν να δούμε τι είναι δυνατό να επιτευχθεί και τι είναι εφικτό να πετύχουμε. Γι' αυτό προσπαθούμε να διερευνήσουμε το πώς θα ήταν δυνατόν να επιστραφούν στο Αζερβαϊτζάν τα κατεχόμενα εδάφη με έναν αποδεκτό τρόπο για την ασφάλεια και για την αυτοδιάθεση του λαού των πολιτών στον εγκόρνο Καραμπάχα. Και δεύτερον, το πώς μπορούμε να παράσουμε μια ασφάλεια στην, στο επίπεδο της αυτοδιάθεση ε, με έναν αποδεκτό τρόπο για το Αζερβαϊτζάν, προτείνοντας να προτείνουμε σε μια μεταγενέστερη φάση την οριστική απόφαση που θα ληφθεί μέσω ψηφοφορίας ούτω ώστε να επιληθεί το θέμα του τελικού στάτους του Ναγκόρνο Καραμπάχα. Ε, το μοντέλο αυτό το 2005-2006 και το προτείναμε όπως είπα ήδη στη Μαδρίτη σαν ε, σε μια γραπτή μορφή ε, είναι οι λεγόμενες αρχές της Μαδρίτης, ε, αποτελούνται από 4-5 σελίδες, 14 αρχές, συν ένα νομικό προήμιο και αυτά έγιναν θετικά δεκτά το 2008 από τις δύο πλευρές. Η διεθνής ε, αναγνώριση για την ανεξαρτησία του Κόσοβο δυστυχώς προκάλεσε πολλές ανησυχίες στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και όλο το 2008 είχαμε πολλές δυσκολίες με το Αζερβαϊτζάν. Ωστόσο το 2009 κάναμε σημαντικές προόδους και είμαστε πολύ κοντά σε μια επίλυση. Οι τρεις πρόεδροι, συμπρόεδροι ανέλαβαν την ευθύνη να δημοσιοποιήσουν στην δήλωση της Λακίλα την ουσία της συμφωνίας την οποία προτείνουμε. Αυτή η δήλωση Λακίλα είναι η έκτη σημαντική πρόταση την οποία ανέφερε ο Μπομπ Μπράτκε και αποτελεί μία σύνοψη των 14 σημείων ε, αρχών της Μαδρίτης. Το 2009 ε, θεωρήσαμε ότι πραγματικά μπορέσαμε να προχωρήσουμε σημαντικά και το 2009 η δήλωση της Μόσχας στη δήλωση της Μόσχας οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα πρέπει να θα πρέπει να υπάρξει ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης μια ειρηνική λύση, η οποία να είναι νομικά δεσμευτική και η οποία να βασίζεται στους διεθνούς κανόνες. Και ευτυχώς οι Ρώσοι, όταν οι Αρμένοι είπαν ότι δέχονται το κείμενο αυτό του, του 2008 τη νέα διατύπωση η νέα διατύπωση η οποία παρουσιάστηκε το 2010 θεωρήσαμε ότι θα ήταν επαναστατική. Αλλά δυστυχώς την εποχή εκείνη μόνο το Αζερβαϊτζάν συμφώνησε με το κείμενο αυτό. Και έκτοτε εργαζόμαστε σε διάφορα επίπεδα ε, από την σαν της κορυφή στο Σότσι όπου εκεί κάναμε κάποια πρόοδο ούτως ώστε και ελπίζουμε πρόοδος αυτή να υπάρξει σε γραπτή μορφή στο εγγύς μέλλον. Εν πάση περιπτώσει ε, φτάνουμε στο τέλος δηλαδή του τρίτου γύρου. Δηλαδή είτε θα είναι πολύ σύντομα δυνατό να εφαρμόσουμε αυτό το μοντέλο το οποίο προτάθηκε το 2007 και διευκρινίστηκε στη συνέχεια ή εάν όχι θα είναι αναγκαίο να εξερευνήσουμε ένα νέο μοντέλο. Δεύτερο σημείο γιατί είναι πολύ προσαρμοσμένο το παρόν επίπεδο των διαπραγματεύσεων. Ε, καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι κάθε μια από τις τρεις χώρες έχει μια, ένα μακρόχρονο και διαφορετικό συμφέρον αλλά η αρμένη της Διαποσποράς στη Ρωσία είναι εξαιρετικά ισχυρή. Η δεύτερη είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τρίτη στη Γαλλία. Το μοντέλο αυτό είναι ενδεδειγμένο ούτω ώστε να παράσχει μέσα των διαμεσολαβητών ένα υψηλό επίπεδο εμπιστευτικότητας η οποία απαιτείται και από τις δύο πλευρές. Και θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, συζητούμε με την ε, Προεδρία και μας συνδράμει ένα πρόσωπο από το Υπουργείο. Δεύτερον, είναι δεδειγμένο για να παράσχει μια συνέχεια. Ο Ρώσος προκάτοχος του τωρινού Ρώσου διαμεσολαβητή Ε, ήταν επικεφαλής ομάδας για 6 χρόνια. Εγώ είμαι στο αξίωμα αυτό εδώ και 6,5 χρόνια. Τέλος, η ομάδα αυτή είναι αρκετά ευέλικτη και αντιδρά πολύ γρήγορα, με μεγάλη ταχύτητα. Και θα ήθελα να σας δώσω μερικά παραδείγματα μετά τη σύγκρουση μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας, όλοι πίστευαν ότι είχε πεθάνει πλέον η ομάδα του Μίνσκ. Ακόμα κατά την περίοδο που οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ρωσία δεν μπορούσαν να συνεργαστούν, η Γαλλία συνέχισε τις εργασίες της εκ και των δύο. Τελικά το σύστημα αυτό είναι αποτελεσματικό γιατί επιτρέπει ταχείες αποφάσεις, σκληρές αποφάσεις, ε, πολύ γρήγορα. Ε, μερικά παραδείγματα. Το 2008 μεγάλες συγκρούσεις στην γραμμή της ανακοχής. πιο σημαντικές, ήταν οι πιο σημαντικές ε, συγκρούσεις συγγνώμη, από την εποχή της ανακοχής, εγχειρίας. Αλλά ο Αμερικανός συμπρόεδρος, ο οποίος ήταν στην εποχή εκείνη, ε, μπόρεσε να παράσχει τις ε, ενδεδειγμένες αντιδράσεις και να αποφύγει μια κλιμάκωση. Τέλος, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίλυση αυτής της σύγκρουσης είναι απολύτως καθοριστικός. Αλλά προσλαμβάνει διάφορες μορφές που είναι προσαρμοσμένες στις διαδοχικές φάσεις της διαθέτησης. Ε, στην παρούσα φάση όπου η, η διευθέτηση θα πρέπει να είναι εμπιστευτική. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστικός στην προετοιμασία της κοινωνίας των ε, πολιτών. Η προαγωγή της ε, δημοκρατίας, εάν δεν υλοποιηθεί, δεν θα είναι δυνατόν οι δύο πρόεδροι δεν θα μπορέσουν να περάσουν από τους λαούς τους την ενδεχόμενη συμφωνία. Συνεπώς λοιπόν αυτό είναι ένα καθοριστικό στοιχείο. Ε, χρησιμοποιώντας όλους τους μοχλούς, όπως είναι η PCA, τα προγράμματα δράσης, η πολιτική γειτονία, μοχλή, που δεν έχουν άλλοι διεθνείς παράγοντες. Μεσοπρόθεσμα η η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίξει σημαντικό ρόλο προς τη διαθέτηση της σύγκρουσης συνεισφέροντας στις ε, παγκόσμιες προσπάθειες όσον αφορά την ανοικοδόμηση και τη συμμετοχή ίσως ορισμένων ε, μελών στις ε, διεθνείς ειρηνευτικές δυνάμεις. Από την άλλη, ε, θα, πρέπει να, θα μας πρέπει να συσταθούν κάποιο διεθνές ε, όργανο όπως ε, για παράδειγμα στη Βοσνία το Συμβούλιο Επέντρωσης της Ειρήνης ούτως ώστε να κινητοποιηθούν όλες οι διεθνείς προσπάθειες συμπεριλαμβάνοντας αυτές των τριών χωρών που έχουν τη συμπροεδρία καθώς και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των χωρών δωρητών, ε, που θα είναι αναγκαίο να κινητοποιηθούν, γιατί η προσπάθεια που θα καταβληθεί είναι τεράστια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Φασιέ. Ο κύριος Κάσπερτσεκ, εκπρόσωπος της ε, Προεδρίας, εναλλασσόμενης Προεδρίας του ΟΑΣΕ όχι πάνω από πέντε λεπτά παρακαλώ, δεν τα πετύχατε εσείς, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω τώρα βλέποντας το ρολόι σας να προσαρμόσετε τον χρόνο μιλία σας με, όπως και κάποια τους προηγούμενους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές. Έχετε μια γενική εικόνα για το τι γίνεται με τη διαδικασία επίλυση των ε, συγκρούσεων και εγώ θέλω να σα συμπλώσω αυτό το κατακούτελο για να δούμε λίγο τι γίνεται όσον αφορά την εντολή ε, για τη δραστηριότητα του μόνιμου εκπροσώπου για να δείτε τι γίνεται ή στο μέτωπο. Ε, Ακριβώ όπω μπορέσαμε να διαπιστώσουμε. Έχουμε τον μόνιμο εκπρόσωπο τον Αύγουστο του 1995 και εγώ τον Ιούλιο του 1996 διορίστηκα αυτή τη θέση και επίση έλαβα από τι επόμενε Προεδρίε, παρά τι εντολίε μου έχουμε ε, έδρα το ε, Μπακού και το Γερεβάν και το την, ε, την, την Τυφλίδα αλλά και τον Αγγόνο Καραμπάχ με το προσωπικό μας κατόπιν των διαπραγματεύσεων έχουμε δει το ότι έχουμε τρεις οι οποίοι πηγαίνουν από τη μία έδρα στην άλλη έχουμε δύο, διεθνείς, δύο μέλη διεθνών αποστολών στην Τυφλίδα η, και η εντολή ε, καλύπτεται τα εξής όσον δραστηριότητα πρώτα πρώτα να βοηθήσουμε το τα εμπλεκόμενα μέρη ε, να απειλήσουν τη διαφορά και όπως ε, θα φαντάζετε ε, προσπαθούμε να συναντηθούμε σε τακτικά διαστήματα με το εμπλεκόμενα μέρη με αρχηγούς κρατών, με υπουργούς να έχουν η όλη ενημέρωση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά τώρα τα λεγόμενα μέρη. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις σχέσεις των μερών. Συνέχεια πηγαίνουμε επί τόπου ε, και τον Οκτώβριο πήγαμε και καλύψαμε 1500 χιλιόμετρα σε τρεις ε, περιπτώσεις μπορούσα να διαπιστώσω τι γίνεται και πιο πρόσφατα πήγα ε, την περασμένη εβδομάδα βοηθούμε όλα τα μέρη. Το πιο σημαντικό είναι το να έχουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη και επίσης να μπορέσουμε να μειώσουμε το μίσο στην προκατάληψη μεταξύ των δύο λαών, να μπορέσουμε και τις δύο πλευρές να τις βοηθήσουμε λέοντάς του ότι αυτό είναι το επιθυμητό και ότι θα πρέπει να προβούν σε συμβασμού για να προχωρήσουν. Ε, οπότε έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουν μειωθεί οι απώλειες και επίσης με αυτόν τον τρόπο ε, μπορούμε να έχουμε καλύτερη ατμόσφαιρα για τι διαπραγματεύσει. Η εντολή μου μου επέτρεψε σε διαφορετικά διαστήματα να διευκολύνω και κάποια ε, πολιτικά ε, πολιτικές κινήσεις και τις δύο πλευρές διαφόρων κινημάτων. Έχουμε και στρατιωτικά μέτρα που τα προωθούν οι στρατιωτικοί κύκλοι, οικονομικά μέτρα, περιβαλλοντικά και τα ΜΜΕ. Οι ύστερες εξελίξεις ε, έδειξαν ότι χρειάζονται περισσότερα μέτρα και κυρίως από το πλευρά του Αζερμπαϊτζάν και δεν μπορούμε να έχουμε οικοδόμηση εμπιστοσύνη άπαξ και παραμένει η κατοχή των του, του, εδαφών του Αζερμπαϊτζάν. Επομένως, μόνο όταν έχουμε ένα μέτωπο θεωρούν αυτοί ότι μπορούν να συνεχίσουν τι διαπραγματεύσεις. Έχουμε μια γραμμή επαφής 650 χιλιόμετρων. Αυτό όμως γίνεται μόνο αν έχουμε από τα εμπλεκόμενα μέρη εμπιστοσύνη. Το γραφείο μας είναι η μόνη διεθνή παρουσία που έχει πρόσβαση στο, στο μέτωπο. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει 12 ε, ασκήσεις παρακολούθησης. Δύο κάνουμε συνήθως μηνιαίως και προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε τακτικά για την κατάσταση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κάποια συμβάντα όπως ε, και μία συμπλοκή με, με τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες ε, είναι δυνατόν στα εμπλεκόμενα μέρη να δίνω τη πιστή εικόνα των όσων έγιναν και έτσι μην έχουμε κλιμάκωση. Επίσης τώρα θα πρέπει να δούμε και τα θέματα τα ανθρωπιστικά. Ε, θα πρέπει να μην έχουμε ένταση, μην έχουμε τελικά επιδείνωση του, τη, της ζωής των, των ε, λαών του ενός και του άλλου αλλά θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη και εμείς επομένως έχουμε στενή επαφή με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Με τον Ερυθρό Σταυρό και αυτό αφορά τους πολίτες, τον ομοχοπληθισμό, κρατουμένους και ασχολούμαι με αυτό τα τελευταία 15 χρόνια. Έγιναν διάφορες παραδόσεις, απελευθερώσεις στο Αστραχάν, στο Σότσι, κατόπιν ε, συμφωνίας των Πρόεδρων και παρουσία του κ. Μεντβέντεφ. Έγιναν τις κορυφές του Σότσι. Οπότε διερευνήσαμε κατά πόσο είναι δυνατόν να διερευνήσουμε το αν μπορούμε να έχουμε κάποια κάθε εικόνα από τα επεισόδια στο μέτωπο. Τέλος όπως προβλέπει η εντολή αναφέρω τις εξελίξεις και τις κινήσεις εποπτείας. Επίσης ενημερώνω όσους εμπλέκονται όσους ενδιαφέρονται όπως τις, τους φορείς κοινωνίας των πολιτών. τώρα από Πέρσι έχουμε σταθεροποίηση. Βέβαια συνεχίζονται οι πυροβολισμοί, οι τραυματίες στο μέτωπο. Όμως δεν επιδεινώθηκε η κατάσταση. Οπότε έχουμε 17 νεκρούς στη γραμμή επαφή, στα σύνορα τέλο πάντων, το πρώτο πεντάμινο φέτο. Και 18 τραυματίες. Όμως είχαμε 35 νεκρούς πέρσι και 52 τραυματίε συνολικά για το 2010. Ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε τα περισσότερα νούμερα. Εάν προχωρήσουν οι πραγματεύσεις θα μειωθούν και οι απώλειες. Θα έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε σε μετακόδομες εμπιστοσύνη. Αυτά όσον αφορά τον ε, επίσημο εκπρόσωπο, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες γιατί νομίζω ότι έχουμε μια οπτική γωνία που δεν έχει κανείς άλλος εμείς ε, και επί τόπου. Ευχαριστούμε για την συνεχή, συνεπή σα στήριξη για μένα και για την ε, ομάδα συνεργατών. Και εδώ μας έχετε βοηθήσει και το Συμβούλιο, οπότε πρόθυμα απαντήσω τυχόν ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πέτρη. Ο Πέτερ Σένεμπι, τέος ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Κάφκασο. Όχι πάνω από πέντε λεπτά παρακαλώ. Πρέπει να συμβουλεύεστε το ρολόι για να σας καθοδηγήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την πρόσκλησή σας σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση. Ξεκινήσω λέγοντας ότι θα μιλήσω σε προσωπική βάση γιατί δεν έχω πλέον τη θέση του αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή του Νοτιού Καυκάσου. Θεωρώ ότι αυτή η συνάντηση είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτήν την τόσο σημαντική αλλά και άγνωστη σύραξη και τη σημασία που έχει για την Ευρώπη. Να πω εκ των προτέρων ότι η σύγκρουση του Ναμπόρνο Καραμπάχ είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης στο Νότιο Κάυκασο και στο σύνολο περίπου της ανατολικής γειτονική ζώνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Νακόρνο Καραμπάχ είναι βασική πηγή ανασφάλειας στην περιοχή εξίσου σημαντική και σοβαρή με την σύγκρουση στη Γεωργία η οποία προς το παρόν ελέγχεται βέβαια. Γιατί είναι σημαντικό το θέμα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο προκαλεί ένα αγώνα εξοπλισμών σε μια ευαίσθητη περιοχή, κάτι το οποίο δημιουργεί περισσότερα προβλήματα για πιθανή χρήση βίας στην περιοχή δημιουργεί προβλήματα και σε περιοχές, στην ευρύτερη περιοχή, σαν παράδειγμα στους ενεργειακούς διαδρόμους, στον ρόλο της Τουρκίας. Δημιουργεί επίσης προβλήματα σχετικά με τις προσπάθειες μείωσης του κόστους προμήθειας της ενέργειας για πάρα πολλές χώρες. Είναι ένας παράγων ανασφάλειας η Γεωργία φοβάται ότι αν υπάρχει μια κάποια σύραξη τότε θα υποστεί και η Γεωργία τις πιέσεις ε, στην περιοχή. Το θέμα αν ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι πράγματι δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι ο φόβος τον οποίο νιώθουν οι Γεωργιανοί. Αυτό έχει σημασία. Γενικότερα, η σύγκρουση στον Αγκόρνο Καραμπά είναι μια ολοένα αυξανόμενη απειλή ε, στα οικονομικά συμφέροντα και τα πολιτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης γενικότερα στην περιοχή του Νοτιού Καυκάσου. Ποια είναι άραγε τα εμπόδια για την ύπαρξη μιας κάποιας λύσης μέχρι τώρα. Καταρχάς, η έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Η σχετική έλλειψη ενδιαφέροντος επίσης της δύση είναι κάτι το οποίο έχει παίξει ένα αρκετά σημαντικό παράγοντα, ιδιαίτερα μέχρι πρόσφατα. Αυτό άρχισε να αλλάζει βέβαια με τους ηγέτες των τριών χωρών που εκπροσωπούνται στη συμπροεδρία της ομάδας του Μίνσκ οι τελευταίες δηλώσεις, τα τελευταία χρόνια μάλλον, οι δηλώσεις αυτής της ομάδας, των χωρών αυτών, στα πλαίσια της ομάδας του Μίνσκ και στα πλαίσια της ομάδας των 8, δείχνουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς αυτών των χωρών και των περιοχών. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει την κατάσταση. Πολλά ακούστηκαν γύρω από αυτό ήδη. Νομίζω ότι μια καλή αρχή θα ήταν να ε, υπάρξει, να στρέψουν την προσοχή τους στο τι έχει συμβεί στην περιοχή και στις εργασίες του Συμβουλίου επίσης. Ελπίσεις μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει σε επίπεδο πόρων για την βελτίωση της ασφάλειας στη γραμμή επαφής των δύο χωρών αυτών, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης κτλ αναφέρθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προωθήσει και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Κάποια από αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη από το πακέτο ΟΑΣΕ Αυτά μπορούν να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο σε, στον τομέα των πολιτιστικών, στον τομέα της συνεργασίας των υπηρεσιών καθολικού συμφέροντος, των προσπαθειών συνεργασίας των χωρών αυτών στον τομέα της απόσύψης και περισυλλογής, περισυλλογής των ναρκών ο ρόλος των μέσων επίσης και η αποφυγή κλισέ είναι και αυτός ένας ρόλος που θα μπορούσε να βοηθήσει. Ε, για να υπάρξει εμπιστοσύνη πρέπει να υπάρξουν και διαβεβαιώσεις από πλευράς της ηγεσία των ε, δύο χωρών εδώ απαιτείται να υπάρξουν περισσότερες επισκέψεις ε, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες της περιοχής, οι οποίες θα επηρεάσουν τις αρχές των χωρών αυτών. Η ανατολική γειτονία, η πολιτική ανατολικής γειτονίας μπορεί επίσης να παίξει σημαντικό ρόλο για την προώθηση των ε, μορφών συνεργασίας Σαν παράδειγμα θα μπορούσαμε να δώσουμε συστάσεις για την ανάπτυξη των υποδομών στην περιοχή μετά την τελική ρύθμιση που είναι ένα θα έλεγα είναι ένα σε εισαγωγικά καρότο το οποίο θα προσελκύσει, θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των εμπλεκομένων μερών. Συμπερασματικά λοιπόν να πω ότι Όσο επιταχύνονται οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτήν την όχι και τόσο γνωστή αλλά σημαντική απειλή θα πρέπει να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει καλύτερα την ανθρωπιστική κατάσταση και να μην αγνοήσουμε το ότι ε, έχουμε ακόμα μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία μπροστά μας όχι μόνο για την υπογραφή της βασικής συμφωνίας αλλά και τις θέσεις εφαρμογή των αποφάσεών της. Νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξει τον Αγκόρνο Καραμπά σε μια ευρύτερη εικόνα για την περιοχή και να προωθήσουμε τους τρόπους συνεργασίας συνολικά με την περιοχή. Το Ναγκόρνο Καραμπά παίζει ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό ρόλο σε επίπεδο στρατηγικών μεταφορών. Έχει ένα διάδρομο μεταφορικό πολύ τιμό ε, για τις χώρες της περιοχής και θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν καταλήτης και κινητήρας για την βελτίωση των συνθήκων επίλυσης του προβλήματος. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέσβη. Κλείνουμε την παρουσίαση των ε, ε, μιλητών με την παρουσίαση του κυρίου Λάιτσκα, ο οποίος θα μας πει την άποψή του για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε το ρολόι σας κύριε Λάιτσκα. Σας παρακαλώ μην το αγνοήσετε και μην ξεπεράσετε τα πέντε λεπτά. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα το κάνετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή είμαι ο μόνος εκπρόσωπος των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, θα εστιάσω την παρέμβασή μου στο τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζοντας την επίλυση της σύγκρουσης των Αγκώνων Καραμπάχα. Θα είναι, είναι διατεθειμένη να προβεί σε διαπραγματεύσεις. Τον Αγκώνο Καραμπάχα είναι το, η μόνη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην περιοχή αυτή ε, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρεμβαίνει άμεσα. Θέλουμε μια πιο ενεργό παρέμβαση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίλυση της σύγκρουση. Ωστόσο έχουμε επίγνωση ότι αλλαγέ στο παρόν επίπεδο των διαπραγματεύσεων, σε, αυτό σε αυτή την ευαίσθητη φάση όπου ε, διαπραγματεύονται ακόμα τις αρχές τις βασικές αρχές δεν θα οδηγήσουν σε μία επίλυση. Γι' αυτό βλέπουμε τη δυνατότητα επανέμβαση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποστήριξη ε, των προσπαθειών για την επίλυση της ε, κρίσης ε, εκτός του υπάρχοντος πλαισίου. Ωστόσο θα θέλαμε να συγχαρούμε το έργο της ομάδας του Μίνσκ που βασίζεται σε σημαντική εμπειρία για την πρόληψη των συγκρούσεων και την επίλυση των συγκρούσεων. Ένας από τους βασικούς στόχους της ε, ε, είπα εκπροσώπου που θα διοριστεί το Σεπτέμβριο αυτού του έτους θα είναι να συνεισφέρει σε μια πετυχημένη επίλυση των συγκρούσεων στην περιοχή και στον Αγκόρνο Καραμπάχα. Θα συμβάλλει λοιπόν στην ε, ενίσχυση του επίπεδου πληροφόρηση όσον αφορά την επίλυση της, σύγκρουσης. Και αυτό σε συνεργασία με την Προεδρία του Μίνσκ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει ένα πιο ενεργό πολιτικό ρόλο μέσω ενισχυμένου διαλόγου με τη συμπροεδρία της ομάδας του Μίνσκ και με άλλου αδικού εταίρου όπω είναι η Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περάσει ισχυρά μηνύματα καταδικάζοντα τη χρήση βία και να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι μόνο μια ειρηνική λύση μπορεί να γίνει υποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να πιέζει και τι δύο πλευρέ στη γραμμή επαφή των δύο χωρών, ε, θεωρώντα την είναι δικαιολόγητη χρήση βία και η θανάτωση πολιτών. Ε, θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στη γραμμή επαφής των δύο χωρών. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να συνεχίσει και να ενισχύσει την υποστήριξή της για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και για την ε, εφαρμογή της ε, και για την, ε, για την επιστροφή των προσφύγων. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στη διαθέτηση της λύσης με 2 εκατομμύρια ευρώ οικονομική υποστήριξη προς μη κυβερνητικού οργανισμούς, οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η χρηματοδότηση είναι ισχνή, αλλά είναι σημαντική για να δημιουργήσει πιο μετριοπαθείς στάσεις και από τις δύο πλευρές μεταξύ νέων πολιτών και παραγόντων που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη ούτως ώστε να ενισχυθεί η δέσμευση στην κατεύθυνση διαθέτηση της κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράσχει σημαντική συνδρομή για την υποστήριξη της δημοκρατική διαδικασία και της ένωμης τάξη στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονία. Επιπρόσθετα, η εντατικοποίηση των σχέσεών μα με αυτέ τι χώρε μέσω των συμφωνιών σύνδεση έχουν σαν στόχο να φέρουν τι χώρε αυτές πιο κοντά στην Ευρώπη από πολιτική και οικονομική άποψη και να συμβάλλουν σε μια πιο ανοιχτή δημοκρατία και στις δύο αυτές κοινωνίες. Θα πρέπει να είναι πιο προετοιμασμένε, να αναμένουν μια ειρηνική διευθέτηση τη σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχα ε, η, ειρηνική, η συμφωνία ειρήνης θα αλλάξει την περιοχή αυτή σημαντικά και θα δημιουργήσει πολλές νέες ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή επιληθεί η σύγκρουση πρόκειται να βοηθήσει στην εφαρμογή. Ε, και, το γεγονός είναι ότι μη επιλημμένες συγκρούσεις στην περιοχή αυτή έχουν αρνητική επίπτωση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό η σύγκρουση στον Αγκόρνο Καραμπάχ είναι και δικό μας πρόβλημα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαδραματίσει ένα ρόλο που να είναι σε πλήρη συμφωνία με την παγκόσμια ευθύνη μας, με την ευθύνη μας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σας ευχαριστώ και για την συντομία με την οποία εκφραστήκατε κύριε Λέτσκα. Πρώτος ομιλητής από πλευράς μας είναι ο κύριος Κυριλόφ, συγητής για τον Νότιο Κάφκασο της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ δύο λεπτά αυτή τη φορά, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εάν πρόκειται για ένα δίλεπτο θα πρέπει να παραλείψω πολλά από εκείνα τα οποία θα σας ε, έλεγα πάντως. Το βασικό είναι ότι τα τελευταία μαντάτα έδειξαν ότι έδειξαν άλλα πράγματα. Τα, τα, τα, τα, τα, οι φήμες είναι διαφορετικές από όσα μας λέτε εσείς, δεν τα ξέρετε εσείς. Άλλα λέει Μόσχα, εμείς είμαστε εδώ. Τι γίνεται. Δεν άκουσα τίποτα από αυτά που ήξερα από εσά. Αυτό τι μου λέει. Ότι θα πρέπει να εξαρτώμεθα από αυτά που μας λένε οι Ρώσοι. Οπότε, η ερώτηση προς τους δύο πρέσβες είναι είστε πεπισμένοι 100% ότι πραγματικά ο κ. Μέντβεντεφ θέλει να αποσπάσει κάποια αποτελέσματα διότι κατά τη γνώμη μου μετά από περίπου μια εικοσαετία που υπάρχει αυτή η ομάδα ε, βλέπουμε ότι μάλλον επικίνδυνα έχουν γίνει τα πράγματα. Παρά το ότι ε, ναι, λένε ότι το, το επεισόδιο το, το, το, το παγωμένο ξαναζεστάθηκε. Ο, δεν, δεν θέλω να γίνω τώρα απολογητής της Ρωσίας, απλώς θα σας πω ότι είναι επικίνδυνο κανείς να έχει τα βγάσει ένα καλάθι δύσκολα να πάρουμε αποτελέσματα. Φυσικά και εδώ και πολύ καιρό ε, πέπρωτε να παίξει σημαντικό ρόλο η Ρωσία και επικοδομητικό μπορεί να είναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι που ενδιαφέρονται. Ε, ε, η υπόθεση του Ναμπούκο, το έργο αυτό και κάποιοι στη Ρωσία θεωρούν ότι η παράταση της σύγκρουσης δεν, δεν Επομένω. Αυτό μόνο προθέσω θα σα ρωτήσω. πάνω στο πιο σημαντικό είναι η δεύτερη ερώτηση που έχω να θέσω. Ευχαριστώ, ξέρω με πρέσβη. Αλλά από αυτό το οποίο μα είπατε, πάνω να πει ότι δεν υπολογίζεται και πολύ τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες την Ευρώπη. Μα λέτε για προπαρασκευή απλά της κοινωνίας των πολιτών και για τις δύο χώρες. το ψήφισμά μας πριν από ένα χρόνο ζήταγε να παίξει πιο δυναμικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, αν γίνει το, το μπάμ όπως θέλουμε και από τη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τα μαζέψει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καλύψει τον κόσμο που θα υποφέρει, τους πρόσφυγες κλπ. κλπ. Η καυτή πατάτα στα δικά μας χέρια θα έρθει. Ευχαριστώ κύριε Κυριλόφ. Η κυρία Γέτεν Μάκη, η συγγήτρια για τις ε, σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν. Δύο λεπτά κυρία Γέτεν Μάκη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που πήρατε μέρος σε αυτήν την τόσο επίκαιρη και χρήσιμη συνάντηση. Όπως ακούσαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει ένα μεγαλύτερο ρόλο στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν και δεν είμαι πεπισμένη ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει στα πλαίσια των υπαρχουσών δομών και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει και μια ξεκάθαρη στρατηγική για το πώς να εφαρμόσει την πολιτική πρόληψη συγκρούσεων την οποία έχει. Θα ήθελα ταυτόχρονα να πω ότι μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση Τι πιστεύετε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα ειδικό αντιπρόσωπο στην περιοχή, ο οποίος να συντονίζει τις προσπάθειές της. Είπατε ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε την κοινωνία των πολιτών. Τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε, πώς θα το κάνουμε και μέχρι τώρα έχουμε κάνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα τελευταίο, σαν εισηγήτρια της ΑΦΕΤ για τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Αφγανιστάν, με το Αζερμπαϊτζάν, συγγνώμη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές όσο περισσότερο γίνεται, όχι μόνο για να φέρουμε πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις χώρες του Νοτιού Καυκάσου αλλά να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να συνεργαστούν και μεταξύ τους. Και αυτό είναι δύσκολο γιατί ακούσαμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης Αντίθετα θα πρέπει εμείς ε, τις ε, ε, λύσεις αυτές να τις προωθήσουμε βοηθώντας την επίλυση την πολιτική του προβλήματος. Γι' αυτό λέω τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ κύριε Γέτεμπάκη. Ο κύριος Κασουλίδης δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τους ομιλητές, τους εκπροσώπους της ομάδας του Μίνσκ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη. Η πρώτη αφορά τις έξι βασικές αρχές. Μία από τις βασικές αρχές αναφέρεται στον μελλοντικό καθορισμό του νομικού καθεστώτος του Ναγκόρνο Καραμπάχ μέσω μιας νομικά δεσμευτικής έκφρασης ε, της επιθυμίας της κάθε χώρας. Παρ' όλα αυτά ακούμε κάποιες δηλώσεις του Προέδρου Αλίεφ, ο οποίος λέει ότι η βασική προϋπόθεση για να δεχθεί είναι ότι δεν θα δώσει ούτε αυτονομία στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάκ στο εσωτερικό της ε, εθνικής κυριαρχίας του Αζερβαϊτζάν. Το δεύτερο θέμα αφορά κάποια ανησυχία που υπάρχει εδώ στο Κοινοβούλιο για την κατάσταση επιτόπου σχετικά με την κούρσα των αγώνα των εξοπλισμών, κάποιες συγκρούσεις, κάποιες στρατιωτικές ασκήσεις και μια πολεμοχαρή ρητορική ότι θα επελευθερώσουμε τον Αγκόρνο Καραμπάχ μέσω των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Αγκόρνο Καραμπάχ. Ενδιαφέρον εδώ είναι ότι οι δύο ηγέτες του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας έχουν ανάγκη την υποστήριξη του λαού τους για να οδηγήσουν ε, σε μία λύση η οποία έτσι και αλλιώς θα είναι οδυνηρή και για τις δύο πλευρές. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μάθω τον Αγκόρνο Παραμπάχ ε, ε, αυτού καλείται να συνεισφέρει στην επίλυση μιας κάποιας λύσης. Έχει κάποιο ρόλο το Στεπάνακερτ. Ευχαριστώ κύριε Κασουλίδο. Κύριος Προβέρα πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούμε για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Πόλεμος, ανασφάλεια κτλ. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το τι συμβαίνει στον Αγκόρνο Καραμπάχ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ιδιαίτερα και σχετικά με τις δυσκολίες που έχουμε με τη Λευκορωσία βέβαια. Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας υπάρχει ένα σημαντικό θέμα που είναι η ειρηνική συνεργασία των έξι χωρών που συμμετέχουν σε αυτό το πάνελ, στις έξι χώρες ενώ της ανατολικής πλευράς. Είναι προφανές ότι τον Ναγκόρνο Καραμπάχ μέσω μιας υποβόσκουσας σύγκρουσης ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν δεν ικανοποιεί τα βασικά κριτήρια για την δημιουργία σχέσεων στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας και των εταιρικών σχέσεων με την ανατολική αυτή πλευρά των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το status quo λοιπόν σε αυτή τη φάση ε, θα έλεγα ευνοεί την αρμενική κατοχή στην περιοχή και αυτό είναι κάτι το οποίο ανησυχεί την κυβέρνηση του Μπακού και προκαλεί ανησυχίες στον πληθυσμό ε, του Αζερβαϊζάν Γιατί υπάρχει αυτό το καθεστώς κατοχής, είναι μια μόνιμη κατοχή εδώ και αρκετά ε, χρόνια, όχι μόνο μάλιστα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλλά και άλλων επτά επαρχιών. Και αυτό θα έλεγα σιγά σιγά τροποποιεί την πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής. Έχουμε την έλευση προσώπων, ανθρώπων οι οποίοι ταυτίζονται με τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, δηλαδή την Αρμενία, και από την άλλη οι αζερικοί πληθυσμοί του Ναγκόρνο Καραμπάχα διαφεύγουν και έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Αυτή η τροποποίηση λοιπόν, η φιλετική και η εθνοτική της περιοχής θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο δημοψηφίσματος για το μέλλον της περιοχής κάτι το οποίο δεν θα πρέπει νομίζω ε, να ε, μας ε, κάνει να μην το δεχτούμε. Πρέπει να είμαστε τολμηροί και θα πρέπει και οι κυβερνήσεις της περιοχής να το δεχτούν. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε και στο ότι τα σύνορα της περιοχής δεν θα πρέπει να αλλάζουν με ένοπλες παρεμβάσεις. Αν πραγματικά υποχωρήσουμε στο επίπεδο αυτής της αρχής τότε άλλες δύσκολες καταστάσεις όπως στην Γεωργία θα, θα προχωρήσουν σε καταστάσεις δυσβάστακτες. Και ε, στο τέλος αν παραβιαστούν αυτές οι αρχές τότε θα υπάρξουν και άλλες μελλοντικές τέτοιες ενέργειες στο μέλλον που θα δημιουργήσουν πολύ περισσότερα προβλήματα για όλους. Ευχαριστώ τον κύριο Προδέρα. Ο κύριος Βάιγκελ για δύο λεπτά παρακαλώ. Όταν άκουσα τον εισηγητή μου γεννήθηκε η αίσθηση ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιες διπλωματικές προσπάθειες σύμφωνα με την βασική παράδοση. Ξέρετε και εγώ ήμουνα στον ΟΑΣΕ διπλωμάτης πρέσβης 98 με το 2. Όμως τώρα έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα πάρα πολύ ε, επικίνδυνο και προσπαθούμε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα το λύσουμε τον κλασικό τρόπο γιατί ήδη έχουμε κάποιες ε, γενιές διπλωματών εξαιρέτων όπως εσείς που ασχολούνται με το πρόβλημα όμως τελικά όπως είπε ο κύριος Προβέρα βρισκόμαστε μόνο στην αρχή έχουμε αυτήν την de facto νοημοποιημένη, αναγνωρισμένη κατοχή. Δεν είπατε εσείς τίποτα για το διεθνές δίκαιο, το οποίο θα έπρεπε να πριτανεύει. Εσείς μίλησατε με πάρα πολύ καλά λόγια για τη Ρωσία που φυσικά και είναι πρωταγωνιστής στην υπόθεση αυτή. Στηρίζονται από τους Ρώσους οι Αρμένοι στις ενεργείες τους. Και πρόκειται εδώ για ένα τελεσμένο το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Και φυσικά για λόγους πολιτικής και σκοπιμότητας ε, πουλάνε όπλα και στις δύο πλευρές. Επομένως, ας μην είμαστε και τόσο επίοικείς προς τους Ρώσους. Ε, κύριε Λάιτσακ, συμφωνώ. Έχετε τα μέσα το οποία χρειάζεται. Και συμφωνώ ότι είπατε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο της. Τα έχετε αυτά που πρέπει τα όπλα, τα εργαλεία και ναι, εμεί μπορούμε να πιέσουμε έστω και λιγάκι το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία αλλά και τη Ρωσία διότι τουλάχιστον αυτές οι δύο τελευταίες χώρες αληθορίζουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπουν στη βοηθειά της Σα είπα, κάνετε την δουλειά με εσά ε, πάνω από μια εικοσαετία. Φυσικά και μπορούμε να το κάνουμε με περισσότερο ομοτρόπο όμως Όμω κάτι θα πρέπει να, να κάνουμε να σκαρφιστούμε κάτι πιο αποτελεσματικό από την κλασική διπλωματία. Ευχαριστώ κύριε Βάιγκελ. Ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημά μου απευθύνεται προς τον κύριο Λάιτσακ και τον κύριο Ζέμεμπι, στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέγραψαν τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μπορούμε δηλαδή να επηρεάσουμε την διευθέτηση της σύγκρουσης. Το ερώτημά μου αφορά τον στρατιωτικό εξοπλισμό στην περιοχή αυτή. Δεν θα ήταν δυνατό σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία συνεργασίας και εταιρικής σχέσης να συμπεριλάβουμε κάποια κίνητρα τα οποία να συνδέονται με μια ξεκάθαρη μείωση των στρατιωτικών δαπανών. Η κυρία Ιμπρισάγκητς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει διατυπώσει τους στόχους μιας επίλυσης. Και είπαμε ότι η Αρμενία, η Αρμενία συγγνώμη, θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τα κατεχόμενα εδάφη. Οι εκπατρισμένοι θα πρέπει να μπορούν να επιστρέψουν στους, στις αιστείες τους. Και επίσης θα πρέπει να εγγυηθούμε την ε, ασφάλεια, τις συνθήκες ασφάλειας. Το είπε και ο κύριος Λάιτσακ ε, εδώ μπορεί να υποπτεύσει εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το ερώτημά μου είναι γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί και τι μπορούμε να πράξουμε το ώστε επιτέλους να εφαρμοστούν. Το, η κατάσταση ως έχει δεν είναι πλέον αποδεκτή και μπορούμε να συζητούμε Μακρόν για το στάτους του Ναγκόρνο Καραμπάχα αλλά θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο μπορεί να προστατεύσει τις εθνοτικές ε, μειονότητες και να εξασφαλίσει τα σύνορα. Υπάρχουν άλλες ε, αντίστοιχες καταστάσεις στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παράσχει μια λύση. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η καλύτερη εξωτερική πολιτική είναι αυτή η οποία μπορεί να επιτυγχάνει στο επίπεδο της πρόληψης κάποιους στόχους, δηλαδή πριν αναθερμανθεί μια σύγκρουση. Και δεν είναι τυχαίο που εδώ στο Κοινοβούλιο θέτουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Εδώ στην Επιτροπή και στην επόμενη Ολομέλη στο Στρασβούργο, αν δεν απατώμε, θα συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο κάναμε μέχρι στιγμή ω Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καθόλου επαρκέ. Ο κύριο Λάιτσεκ είπε ότι δίνονται σε μη κυβερνητικού οργανισμού 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι ευγενικό, αλλά δεν βρίσκεται από πίσω η πολιτική πίεση που είναι αναγκαία για να αποτρέψει τις δύο πλευρές να εξοπλίζονται και να ε, οδηγούνται στον πόλεμο, στην πολεμική σύραξη. Το ερώτημά μου, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι πολλούνται όπλα από τη Ρωσία στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Θα ήθελα να μου το επικαιρώσετε από τη δική σας πλευρά. Και μετά καλώ την Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταβεί εκεί η κυρία Άστον τόσο στον Μπακού όσο και στο Ριβάν και να καταστήσει σαφές και στις δύο πλευρές ότι από μια ενδεχόμενη σύγκρουση θα υποφεληθεί μόνον η Ρωσία γιατί η Ρωσία είναι αυτή η οποία εξοπλίζει και τις δύο πλευρές. Και μετά το πόλεμο θα παίξει το δικό της ρόλο. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ούτε σόφελος του Αζερβαϊτζάν, ούτε της Αρμενίας, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε και υπέρ των δικών μας ενεργειακών συμφερόντων στην περιοχή. Παρακαλώ λοιπόν να διαβάσετε, να διαμηνήσετε στην κυρία Άστον ότι θα πρέπει να το συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη και με όλο το βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθίσει σαφές και στις δύο πλευρές ποιο είναι το πραγματικό του συμφέρον, δηλαδή να εξεύρουν μια ειρηνική λύση από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαντσμπέργκης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα προς τον κύριο Σάνεμπι και στους αξιότιμους πρέσβεις. Τέλος, η ομάδα Μίνσκ τελικά είναι υπεύθυνη εδώ. Εν σχέση με τα όσα υπόθηκαν για τον Αγκόρνο Καραμπάχ τι θα γίνει αν οδηγηθούμε προς ένα νέο πόλεμο. Η σύγκρουση στον Αγκόρνο ο Καραμπάχ ή ο παγωμένος πόλεμος είναι μια βραδιφλεγής ε, βόμβα η οποία μπορεί να εκραγεί ε, ξαφνικά ή τυχαία. Εάν κάποιος έχει μια, ή αν κάποιος έχει μια πρόθεση να το πράξει. Και αν δούμε την εχθρότητα της ε, Ρωσίας προς την ενοχλητικά ανεξάρτητη Γεωργία και εφόσον όλα τα άλλα άλλες προσπάθειες δεν έδωσαν καρπούς ποια, είναι η άποψη η άποψή, η άποψή σας εάν η Ρωσία και η Αρμενία κινηθούν ε, προς, το, ε, προς μια τέτοια κατεύθυνση. Ο κύριος Λίζεκ για δύο λεπτά. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ κύριε Πρόεδρε για την δυνατότητα που μας δώσατε να ακούσουμε τους φιλοξενούμενους ομιλητές. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπαν και ιδιαίτερα τώρα και μετά από την παρέμβαση του κυρίου Λανσπέργης θα ήθελα να πω ότι εδώ και τρεις εβδομάδες επισκέφθηκα στη Γεωργία σαν εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκεί είχα την δυνατότητα να συνομιλήσω με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και τους κοινοβουλευτικούς και εξοκοινοβουλευτικούς παράγοντες. Και υπήρξε μια ομοφωνία θα έλεγα στο σύνολο των γεωργικών, της γεωργικής πολιτικής τάξης σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί στον Αγκόρνο Καραμπά. Υπάρχει ένας τεράστιος φόβος για την κατάσταση στην περιοχή και για τις υποβόσκουσες αυτές, ε, ε, για την υποβόσκουσα αυτή σύγκρουση στην περιοχή. Ίσως να είναι μια υπερβολή, αλλά από την άλλη πριν πάω στην Γεωργία επισκέφθηκα την Τουρκία και η Τουρκία ανησυχεί ιδιαίτερα για το τι θα συμβεί στον Αγκόρνο Καραμπά. Όπως γνωρίζουμε στην Γεωργία υπάρχει μια αρμενική μειονότητα και υπάρχει και μια αζερική μειονότητα και οι σχέσεις ανάμεσα στις μειονότητες αυτές στην Γεωργία εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ καλές. Όμως υπάρχει δυνητικά θα έλεγα μια δυνατότητα να περάσουν ρωσικές δυνάμεις στην Γεωργία σε περίπτωση σύραξης μέσω της Αρμενίας και αυτό θα δημιουργήσει τρομερά προβλήματα. Λοιπόν δεν έχω να θέσω κάποια ερώτηση, απλά θα ήθελα να σας μεταφέρω το τι πιστεύουν στην περιοχή. Ευχαριστώ κύριε Λίζεκ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο πράγματα. Καταρχήν, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νότιο Κάφκασο μου φαίνεται αντιφατική. Από μία πλευρά η υποστήριξη χωρίς καμία αμφισημία της ραφικής ακερότητας της ε, Γεωργίας ενώ ε, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά όσον αφορά το Αζερβαϊτζάν. Δεν πιστεύετε ότι αυτή αυτά τα δύο μέτρα και σταθμά αποδυναμώνουν την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή αυτή. Και δεύτερον, όσον αφορά την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με αυτή τη σύγκρουση, δεν πιστεύετε ότι θα ήταν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθ' αυτή να συμμετέχει στην ομάδα Μίνσκ. Βεβαίω συμμετέχει η Γαλλία. Η Γαλλία δεν ισούται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι είναι σημαντική γιατί είναι πολύ πιο ουδέτερη. Εξάλλου ακούσαμε ότι οι τρεις εταίροι συμμετέχουν λόγω της σημαντικής αρμενικής διασποράς στις τρεις αυτές χώρες, κάτι που δεν ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι θα ήταν ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μέλος αυτής της ομάδας του Μίνσκ. Σας ευχαριστώ. Κλείνει τη συζήτηση ο κύριος Βένσον για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες που, μου δώσατε, που μας δώσατε. Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας αλλάζει και βλέπουμε τις σχέσεις μεταξύ Αρμενίας, Τουρκίας, Αζερβαϊτζάν και Αζερβαϊτζάν, συγγνώμη, να βρίσκονται επίσης σε μια εξέλιξη. Αλλά ενδεχομένω θα μπορούσαμε να θέσουμε κάποια αιτήματα και προς την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με τη σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχα. Γιατί η Τουρκία ε, της, ε, ενδιαφέρεται επίση αυτή η σύγκρουση λόγω των συνόρων της. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς βλέπετε τη σχέση με την Τουρκία ως προς τη σύγκρουση αυτή. Θα δώσω λοιπόν την ίδια σειρά ε, απάντηση στους ομιλητές. Βέβαια δεν υπήρξαν διευκρινήσεις προς ποιους ε, απευθύνονται οι ερωτήσεις και γι' αυτό εξαρτάται από εσά να μοιράσετε λίγο τα θέματα και εδώ όχι πάνω από 5 λεπτά στο καθένα. Ελπίζω ότι όλοι μαζί να μπορέσετε να δώσετε απαντήσεις. Ο κύριος Μπρέκε παρακαλώ έχει το λόγο πρώτος. Πρέσβης κύριος Μπρέκε. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα αυτά τα θέματα κάποια από τα θέματα αυτά είναι περισσότερα θέματα ενδοκοινοβουλευτικά αλλά θα περιοριστώ στο να σχολιάσω ορισμένα σημεία τα οποία έθεσαν ορισμένοι ε, ομιλητές. Ο Ρώσος Αντιπρόεδρος δεν είναι μαζί μας σήμερα και δεν είναι ρόλος μου να υπερασπιστώ εγώ την Ρωσία. Αλλά δεν συμφωνώ με τα σχόλια που έγιναν ότι αφήνουμε το θέμα αυτό στη φροντίδα μόνο των Ρώσων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε τρεις χώρες να συνεργαστούμε και βασικό μας συμφέρον είναι να μην υπάρξει άλλος πόλεμος. Για όλους μας, για διαφορετικούς ίσως λόγους, ένας άλλος πόλεμος θα είναι μια καταστροφή. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε από κοινού. Εγώ ήμουν παρόν σε πάρα πολλέ συναντήσει με τον Πρόεδρο, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και συνεργαζόμαστε και με τους Ρώσους με διαφάνεια, με έναν τρόπο ο οποίος ίσως μου είναι μοναδικός στα 37-38 χρόνια που είμαι εγώ ε, στο διπλωματικό σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποτέ δεν εργάστηκαν με τέτοιο τρόπο με τους Γάλλους βέβαια και τους Ρώσους συναδέλφους. Είναι μια πράγματι ε, ιδιαίτερη στιγμή γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα, συνεργαζόμαστε και σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε την υπόθεση αυτή στη φροντίδα μόνο των Ρώσων ή οποιονδήποτε άλλον. Έγιναν και ορισμένες αναφορές σε βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και ότι δεν αναφερθήκαμε είπατε στις βασικές αυτές αρχές. Πολλά είναι τα θέματα λόγω χρόνου στα οποία δεν αναφερθήκαμε. Υπάρχει όμως ε, που λέει ότι ε, το να επιλέξουμε μία βασική αρχή του διεθνούς δικαίου όπως την εδαφική ακεραιότητα και να πούμε ότι επί τη βάση αυτής της αρχής θα λύσουμε το πρόβλημα, αυτό δεν αρκεί και οι δύο πλευρές θα σας πούνε ότι οι θέσεις τους βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Συνεπώς δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα το να εμείνουμε στο θέμα του διεθνούς δικαίου. Δεν είναι ο σωστός οδηγός για μας. Και οι δύο πλευρές πιστεύουν ότι οι θέσεις τους βασίζονται στο διεθνές δίκαιο με την αρχή της αυτοδιάθεσης, με την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας, με, κάποιες, με κάποια άρθρα της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών κτλ. Υπάρχουν ε, βασικές αρχές, υπάρχουν δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι, διεθνείς συμβάσεις, συμφωνίες. Εμείς όμως θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα πρακτικά πώς μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε και αυτές τις βασικές αρχές και με βάση αυτές τις αρχές να βρούμε λύσεις πρακτικές τις οποίες να δέχονται όλοι. Το Διεθνές Δίκαιο προφανώς και βοηθάει, μας καθοδηγεί θα έλεγα προς μια σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει αυτές τις αρχές ε, να τις ε, μετατρέψουμε θα έλεγα σε πραγματικότητα. Ευχαριστώ κύριε Μπρέ και ο πρέσβης κύριος Φασιέ έχει το λόγο. Βεβαίως. Επιτρέψτε μια που υπάρχει δερμηνία να σας μιλήσω στην γλώσσα του Μολιέρου αφού κατά πρώτη φάση σας μίλησα στη γλώσσα του Σέξπιρ. Έχουμε εδώ μια σειρά απαντήσεων που πρέπει να δοθούν για να καλύψω ένα τμήμα της, ε, των ερωτησιών σας. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν μιλήσαμε πιο λεπτομερώς για τις επιτυχίες που προσδοκώνται για τις επόμενες εβδομάδες βεβαίως και έχουμε προσδοκίες ε, υφηξημένες όμως ήρθε η ώρα κατά την οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάει κανείς τον ανάσα του και να μην πανηγυρίζει πρόημος Οπότε και εμείς νομίζουμε ότι θα γίνει επιτέλους κάποια πρόοδος μέσα στις εβδομάδες, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θα ήταν δόκιμο το να δημιουργούμε προσδοκίες αδικαιολογήτως. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει κάποιος πάρα πολύ ενημερωμένος σχολιαστής των εξελίξεων ή στον Αγκόνο Καραμπάχ που έχει πει εδώ και πολλά χρόνια ότι τίποτα δεν γίνεται και ότι αδιέξοδο για τι διαπραγματεύσει. Στη συνέχεια είχαμε αυτό το συμπόσιο την εβδομάδα ή στον Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε και ο ΙΕ είπε ότι την επόμενη συνεδρία, την επόμενη συνάντηση θα έχει λυθεί ε, το θέμα ακριβώ, αυτό που έχουμε πει πρέπει να αποφύγουμε. Τώρα έχουμε και το θέμα αυτό που είπε ο κύριο Κύριλοφ, ο άπιστο Θωμά, όμω κάνετε λάθο σε σχέση με την ενημέρωσή μα. Είμαστε κάλλιστα ενημερωμένοι σε σχέση με το τι έγινε προχθέ ή στην Μόσχα και εγώ και ο Αμερικανός ομόλογος ενημερωθήκαμε καθόλου όλες τις λεπτομέρειες από τον ε, Συμπρόεδρο. Όμως θα ήταν ανεύθυνο εμείς εκ των προτέρων να αναγγείλουμε προόδους οι οποίες επιτυγχάνονται τώρα ελπίζοντας ότι θα ολοκληρωθούν τις μέσω επόμενε εβδομάδε. Δεύτερον, τώρα στον πρώτο ρόλο τη Ρωσία και για να συμπληρώσουμε αυτό το οποίο είπε ο Αμερικανό ε, συνάδελφο, η απάντηση είναι καταφατική. Είμαι θαυμασμένη ότι η Ρωσία ε, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την επίλυση τη συγκρούσεω. Και εμεί δεν θεωρούμε ότι είμαστε, όπως είπατε, πάρα πολύ επίοικοι και μαλακοί με την Ρωσία, διότι γνωρίζουμε ότι τι γίνεται στη διαδρομή των διαπραγματεύσεων και ότι ε, ε, ε, ξέρω πολύ καλά τι κάνει η Μόσχα όσον αφορά αυτά τα οποία προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις δηλαδή αυτά που συζητούνται σήμερα είναι αυτά τα οποία ο Ρώσος Υπουργό και συνέχεια ο Ρώσος Πρόεδρος πρόκειται να προσπαθήσουν να αποσπάσουν δηλαδή αφορά την συμφωνία επί της τελευταίας εκδοχής του εγγράφου το οποίο εκπονήθηκε και από τα τρία μέρη και η αρχική του εκδοχή συνετάγει από τον προκάτοχο των συναδέλφων Ρώσου, Αμερικανού και του ομιλούντος επίσης για το ρόλο της Ρωσίας. Δεν πουλάει μόνο η Ρωσία όπλα στα εμπλεκόμενα μέρη. Είναι γνωστά αυτά. Και ξέρετε σίγουρα ότι σήμερα στην Ευρώπη ουδέμια χώρα μπορεί να ρυθμίσει, να ελέγξει, να διαχειριστεί το τι γίνεται με τα drone. Για αυτά, τα drone, τα, τα, τα αναγνωριστικά ε, αεροπλάνα που είναι μη επανδρομένα, τα οποία είτε χρησιμοποιούνται για κάποια χτυπήματα, είτε για κατασκοπία. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά στις 26 έκτου, μέσα δηλαδή σε λίγες ημέρες, ή στην ε, παρέλασε τη στρατιωτική του Μπακού θα προκύψει ότι το Αζερβαϊτζάν έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει ντρόουν στη χώρα. Και πώς θα καταφέραν να φτάσουν σε αυτό το σημείο, μια που γνωρίζουμε ότι είπα και άλλη μια χώρα που γνωρίζετε που ελέγχουν την παραγωγή και ότι επίση Γαλλία και Ενωμένο Βασίλειο στην Ευρώπη προσπαθούν να κάνουν κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Άρα κάποιο άλλο. Κάποιο άλλο. Και όχι η Ρωσία. Βοήθησε το Αζερμπαϊτζάν. Όχι, όχι, όχι και όχι είπα, λέει ο, ο κύριος Μπράτια. Όχι, όχι, δεν, δεν κάναμε τέτοια πράγματα. Euh, ναι, ναι, βεβαίω, βεβαίω και ευχαριστούμε για αυτήν την διευκρίνηση. Euh, ε, ε, Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το ρίσκο σε αυτή την κούρσα των εξοπλισμών σήμερα είναι αυτό το παράλογο υπερβολικό επίπεδο που έχει φτάσει. Μην ξεχνάτε ότι ο στατικός προϋπολογισμός ε, του Αζερμπαϊτζάν αυξήθηκε κατά 20-30% ετησίως εδώ και πολλά χρόνια. Και διπλασιάστηκε φέτος. Δηλαδή, φέτος αυξήθηκε κατά 200% ε, και ο προπολογισμό τους, ο είναι πολύ μεγαλύτερος από τον προπολογισμό των κρατικών το συνολικό της Αρμενίας. Να που εγκυμονείται το κίνδυνο και γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ και να σύμφωνα με αυτό που ο Λάιτσακ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ πάρα πολύ επέμεινε όσον αφορά την μη χρήση βίας ε, προχωρήσαμε στις συμπροτρέψεις χώρες, στην Ντοβίλ, τα είπαμε ότι η χρήση βίας ήδη έχει οδηγήσει στην απαράδεκτη σημερινή κατάσταση και ότι αν προσφύγουν και πάλι στην βία τα εμπλεκόμενα μέρη αυτό θα πρέπει να είναι αντικείμενο δίκη από την κοινότητα. σε σχέση με το εάν παραπέμψαν στο διεθνέ δίκαιο. Δεν, με εκπίσω αυτό το πίπεδο, γιατί εγώ σα είπα για τη διακήρυξη τη Μόσχα, όπου για πρώτη φορά οι συμπρόεδροι ε, ή είπαν ότι θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσει οι δύο πρώτοι των δύο χωρών και ότι όλα αυτά θα πρέπει να εδράζονται ή στις αποφάσεις και αρχέ και τα προβλεπόμενα το διεθνέ δίκαιο και σα έχουμε διανύμει και αυτή την ε, τεκμηρίωση όπου έχουμε αυτή τη διακήρυξη της Θανά, όπου οι χώρες απέσπασαν ε, τη σύμφωνη γνώμη των δύο εμπλεκομένων, ότι δηλαδή η ρύθμιση θα πρέπει να βασίζεται εις τους κανόνες του διεθνούς δικαίου στο χάρτη του ΟΗΕ και στην τελική πράξη του Ελσίνκη. Τώρα, γιατί παρά όλα αυτά τα αξιόλογα ψηφίσματα ακόμα δεν πετύχαμε το στόχο μας. Μα είναι απλό. Γιατί δεν το επιθύμησαν τα δύο μέρη. Και είπαμε ότι η διεθνή διαμεσολάβηση ακόμα δεν οδήγησε σε μια συμφωνία. Μα δεν, είναι δυνατόν ο διεθνή παράγων να, να, να, να φτιάξει τη συμφωνία. Ούτε μπορεί να επιβάλλει τη συμφωνία. Θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι να δεχθούν να συμβαστούν. Όμως, και αυτό τα ξέρω μια που έχω υπηρετήσει στη Γεωργία πριν πάω σε Αρμενία και Ζερμπαϊτζάν, προσπαθώ λοιπόν να θεωρήσω ότι η λέξη συμβασμός δεν υπάρχει στη γλώσσα, στον πολιτισμό, στην κουλτούρα αυτών των χωρών. Επομένως, παραμένει πάρα πολύ σημαντικό το να βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις ε, προσπάθειες της ε, στήριξης της ε, ο κ. Στον και ο κ. Κυρδοφή είπε ότι είμαι πάρα πολύ σχετικό ε, για τον ρόλο τη Ένωση. Αποφασιστικό. C'est donc le rôle que je vois pour l'Union européenne, en particulier euh, dans. Επομένω, πρόκειται για αυτόν τον ιδιαίτερο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ε, πρόθεση τη δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ βασικό και η διαπραγμάτευση είναι σαν ένα τρένο που μπαίνει σε τούνελ σε τούνελ, δηλαδή είναι το τρένο προστατευμένο από την ατμόσφαιρα και όπου δεν έχουμε διαρροές. Όταν όμως βγαίνει από το τούνελ, από τη σύραγγα αυτό το τρένο με κάποιο είδους ρύθμιση, όμως τα τρένα της κοινωνίας των πολιτών βρίσκονται στην ε, αναχώρηση, στην είσοδο του τούνελ και κανένας αρχηγός κράτους δεν, δεν πρόκειται να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, να έχει το πολιτικό θάρρος, να προτείνει στο, στο λαό αυτό το τίτλο το συμβασμό, τη συμφωνία. Τελευταίο τώρα. Όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα εξελιχθεί, είπαμε ότι είναι αποφασιστικό σε όλες τις φάσεις, όμως ε, όσον αφορά αυτό που είπε ο συνάδελφος, ο συμπατριώτης, ε, για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς υποκαθιστά τη Γαλλία, ναι, υπάρχει εδώ ένα θέμα. Αυτό ακριβώς που σας τόνισα. Δηλαδή, την πετυχημένη συνταγή που έχουμε για τις διαπραγματεύσεις εάν είναι καταφατική η απάντηση σε αυτά τα θέματα τότε εντάξει εάν είναι δυνατόν να γίνονται όλα αυτά εμπιστευτικά, εντάξει, να δούμε αν θα γίνει όμως έτσι και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξασφαλίσει αυτή τη συνέχεια στις κινήσεις και μιλώ για το συμπρόδρο το Γάλλο, το Ρώσο, μιλώ εδώ και εξατία, 6,5 χρόνια που είναι οι ίδιοι τότε, αν όλα αυτά γίνουν, πολύ καλά θα γίνουν. Και τώρα τελευταίο, αλλά σημαντικό, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εις θέση να μπορεί να κινητοποιηθεί με τρόπο τόσο ώστε μέσα σε μισή μέρα οι τρεις πρωτεύουσε ε, στρατευθούν ε, ε, για να λύσουν κάτι όπως με αυτό το επεισόδιο που έγινε στο, στο μέτωπο το 2008 γιατί το καταφέραν τότε μέσα σε μισή μέρα περάσανε ε, στο, στο ύψιστο επίπεδο τα μηνύματα στους υπουργούς εθνικής άμυνας και στους προέδρους αυτών των, εάν λοιπόν η απάντηση είναι καταθετική αν μπορούμε να ενεργήσουμε μέσα σε μισή μέρα τότε πρίμα τώρα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα για την άσκηση της πολιτικής μας ε, τότε έχουμε αυτή την διακήρυξη της Ντοβίλ, τη δήλωση της Ντοβίλ που είδατε πόσο δυναμική είναι όσον αφορά το μήνυμα το οποίο ήταν πάρα πολύ στόχοθετημένο ε, και για τις δύο εμπλεκόμενες χώρες τότε, τότε να ξέρετε ότι πήρε μία ώρα για να συνταγεί αυτό το κείμενο από τους τρεις συμπροέδρους ούτε το Κρεμλίνο ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε τα ηλίσια άλλαξαν μια κεραία από αυτό το γράμμα. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορέσει να φτιάξει ένα τέτοιο κείμενο μέσα σε μια ωρίτσα, ε, τότε όντω δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να υποκαταστήσει την Γαλλία η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσει. Ε, Ευχαριστώ κύριε Φασιέ. Το λόγο έχει ο επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Κάσπερτσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν ετέθη κάποια ερώτηση σε σχέση με τη δική μου εντολή. Παρ' όλα αυτά σας έδωσα το λόγο. Αν θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ετέθηκαν κάποια ερωτήματα τα οποία μπορούν να χωριστούν σε κάποιες κατηγορίες. Οι ερωτήσεις του κυρίου Κυρίλοφ, Λαντσπέργκης και άλλους αφορούσαν το ρόλο της Ρωσίας. Και θα έλεγα ότι δεδομένες τις εμπειρίες μου μετά από αρκετά χρόνια ε, σε σχέση με το ρόλο της Ρωσίας στην περιοχή του Νοτιού Καυκάσου θα ήθελα να πω ότι μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία έχει προεξάρχον ενδιαφέρον στην ε, διατήρηση και αποκατάσταση επιρροής στο Νότιο Κάφκασο. Γιατί για δύο δεκαετίες ήταν μάλλον σε αμυντική στάση. Τώρα, σε σχέση με τον Αγκόρνο Καραμπάχ ειδικά, υπάρχουν πολλοί στόχοι που προσπαθεί να πετύχει η Ρωσία. Οι Ρώσοι όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις ε, ξεκίνησαν ε, οι ρωσικές πρωτοβουλίες αμέσως μετά και θέλαν να γνωριστούν σαν θετική δύναμη μετά τον όλεθρο του πολέμου στη Γεωργία. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια ευχή να εκμεταλλευτούν τα ανοιχτά ζητήματα ως μοχλό έναντι της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν, ούτως ώστε να προαχθούν τα οικονομικά ρωσικά συμφέροντα. Και τρίτον, παρόλο που αυτή η υπόθεση δεν ε, τη χάνει της κοινή αποδοχής, πιστεύω ότι η Ρωσία καταλαβαίνει την ανάγκη να δράσει προληπτικά, ώστε να μην ξεφύγει η κατάσταση εντελώς ε, καθώς εξελίσσονται τα συμφέροντα της Ρωσίας γιατί κάτι τέτοιο, αν κλεμακώνονταν η σύγκρουση, αυτό θα ήταν εις βάρος της Ρωσίας. Τώρα, όσον αφορά την ε, δυνατότητα μια ανοιχτή στρατιωτική σύγκρουση να ξεσπάσει ένας τυχαίος πόλεμος. Εδώ πιστεύω ότι έχουμε ένα σοβαρό θέμα όσον αφορά τις αβεβαιότητες τις οποίες ήδη αναφέρθηκα και κάτι τέτοιο θα συμπεριλάμβανε και άλλους εταίρους εκτός από την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν και ασφαλώς θα σήμαινε μία απειλή και ανησυχίες ε, για τους Γεωργιανούς από πολλέ πλευρέ. Όσον αφορά το ρόλο τη Τουρκία, ο κ. Σάνσον έθεσε αυτό το ερώτημα και ο Μύρο Λάιτσεκ μίλησε για αυτό το θέμα για το ρόλο τη Τουρκία. Βεβαίω είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί η Τουρκία σε κάποια περιφερειακή προοπτική την οποία θα πρέπει να διατυπώσουμε σε σχέση με τον Νότιο Κάφκασο και που θα προλυάνει το δρόμο για μια επίλυση των συγκρούσεων. Η Τουρκία ε, δεν έπαιξε ένα ρόλο αντίστοιχο με τον ιστορικό της ε, ρόλο και το βάρος της και τη βαρύτητά της. Γιατί ίσως η σύγκρουση στον Αγκόνο Καραμπάχ είναι η πιο σημαντική στην περιοχή. Και δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω εδώ ότι η σύγκρουση του Αγγόρνου Καραμπάχ ήταν πράγματι ο λόγος για τον οποίο η ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας που ελπίζαμε να γίνει πριν από μερικά χρόνια τελικά εκτροχιάστηκε. Η Τουρκία συνεπώς έχει έναν θεμελιώδη ρόλο να παίξει στην επίλυση αυτής της σύγκρουσης. θα που ε, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και ε, οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι ε, συνεχίζουν να προβάλλουν το επιχείρημα ότι θα πρέπει να, συμβεί μια, να γίνει μια ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας που θα δημιουργήσει μια θετική δυναμική και θα συμβάλλει ενδεχομένως στην ε, επίλυση τη σύγκρουση των Αγκόρνου Καραμπάχ. Τώρα όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, ο κύριος Κασουλίδης, ο κύριος Πρισάγκετ, ο κύριος Προβέρο, ο κύριος Βάιγκελ, η κυρία Κιλ Νίλσεν έθεσαν ερωτήματα σε σχέση με αυτό. Η σύντομη απάντησή μου είναι παραπλήσια με αυτή που έδωσε ο κ. Μπράτσκι. Η κάθε σύγκρουση είναι μοναδική. Βεβαίω το διεθνέ δίκαιο θα πρέπει να τηρείται. Αλλά αν μιλούμε για το τι καταλήγει σε μια συμφωνία μετά από μια σύγκρουση. Ε, τελικά είναι μικρός ο ρόλος των ε, διεθνών κανόνων, του διεθνούς δικαίου. Ε, συνήθως πρόκειται για συμφωνίες μεταξύ των πολιτικών μερών που ενέχονται. Ε, τέλος τέθηκε το ερώτημα για, τον, για τη λειτουργία του ειδικού εκπροσώπου, γιατί εγώ είχα αυτό το αξίωμα για πέντε χρόνια και ο Μύρος Λαβλάιτσεκ είπε, εξήγηλε, ότι θα υπάρξει από την 1η Σεπτεμβρίου ένας ειδικό εκπρόσωπος. Και δεδομένης δικής μου εμπειρίας πιστεύω ότι αυτή η σεπτεμβριου ενας ειδικο εκπροσωπος και της δικης μου δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί ενεργά σε θέματα τα οποία ζητούν, ε, προποθέτουν μια ειδική προσοχή. Ε, ε, επαφή υψηλού επίπεδου με τους επικεφαλείς ε, των χωρών στις περιοχές αυτές και το πρόσωπο το οποίο θα καταλάβει αυτό το αξίμα από την 1η Σεπτεμβρίου θα είναι σε θέση πραγματικά να διαδραματίσει ένα ουσιώδη ρόλο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσει τις παρεμβάσεις ο κύριος Λάιτζακ. Θα κάνει και τα τελικά σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πλεονέκτημα το ότι έχουν δώσει, δοθεί περισσότερες απαντήσεις. Θα αναφερθώ και στο ρόλο όμως Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάποια άλλα θέματα. Σχετικά με τον αν θα πρέπει να είναι μέλος της ομάδας του Μίνσκ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές ότι για διάφορες ε, σειράξεις στον κόσμο έχουμε διαφορετικές μορφές. Έχουμε διαφορετική μορφή παρέμβαση στη γεωργία, διαφορετική μορφή στην νηστερία, διαφορετική στο Άνω Καραμπά Θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη μέθοδο. Το να συζητάμε τη μέθοδο και όχι την ουσία των προβλημάτων δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βασιστούμε στις αρχές φυσικά του διεθνούς δικαίου να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και τη δημοκρατία. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Συνδέεται φυσικά το θέμα της Γεωργίας με το θέμα του Άνω Καραμπά, είναι η ίδια περιοχή. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε είναι να συντελέσουμε πρόοδο στην περιοχή γενικότερα και δεύτερον να είμαστε πολύ συγκροτημένοι στις θέσεις που έχουμε και στην προάσπιση των βασικών μας αρχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και τη στρατηγική και τα μέσα. Αναφέρθηκα στα στοιχεία της στρατηγικής μας. Φυσικά όλα θα εξαρτηθούν από την πρόοδο των επαφών Ελπίζω να υπάρξει μια πολιτική ρύθμιση η οποία να ξεκινήσει τουλάχιστον τον επόμενο μήνα και αυτό θα μπορέσει να βελτιώσει και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν υπάρξει εξέλιξη προφανώς θα μπορέσουμε να παρέμβουμε και καλύτερα. Αν υπάρξει στασιμότητα δεν έχουμε πολλές δυνατότητες βελτίωσης της παρουσίας μας θα υπάρξει από το Σεπτέμβριο νέος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή. Αυτό θα προσδώσει μια μεγαλύτερη ορατότητα στην παρουσία μας στην περιοχή. Κάποια σχόλια τώρα για τις συμφωνίες σύνδεσης τις οποίες αναπτύσσουμε με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Πράγματι εγώ πέρασα μια ολόκληρη εβδομάδα στον Μπακού και στον πίληση και στο Γερεβάν Προσπαθούμε για κάθε χώρα να λειτουργήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Κάθε τρόπος όμως θα σέβεται και ε, την πρόοδο σε θέματα επιμέρους, σε θέματα τεχνικά και από την άλλη στον σεβασμό των ευρωπαϊκών αρχών. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τους εταίρους μας να καθορίσουν το επίπεδο των φιλοδοξιών τους, γιατί όσο περισσότερο προχωρούν στις διαπραγματεύσεις, τόσο θα μπορέσουν να ενταχθούν στα ευρωπαϊκά προγράμματα καλύτερα και τόσο περισσότερα χρήματα θα πάρουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προετοιμάζουμε τώρα την Ανατολική Εταιρική Σχέση, τη συνάντηση κορυφής στη Βαρσοβία το Σεπτέμβριο και θα προσπαθήσουμε με κάθε έναν από τους ομιλητές μας ε, να τους εξηγήσουμε τα πλεονεκτήματα για να εμπλακούν ακόμα περισσότερο με τα προγράμματα. Δεν συμφωνώ με το ότι η Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν δεν πληρούν τα κριτήρια. Πρώτον βρισκόμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης των κριτηρίων αυτών και εδώ και δύο εβδομάδες είχαμε εκδώσει θα έλεγα να ορίσουμε τα προβλήματα στις έξι αυτές χώρες και αυτό να το χρησιμοποιήσουμε σαν βάση για περαιτέρω, για περαιτέρω πρόοδο. Δεν υπάρχει λοιπόν δυνατότητα περαιτέρω σύνδεσης ε, των εταιρικών αυτών συνδέσεων με τον Αγκόρνο Καραμπάχ, αλλά παρόλα αυτά είμαστε ξεκάθαροι για την φιλοδοξία που έχουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσουμε τα προβλήματα. Και δεύτερον, όπως σας είπα, για τις αρχές μας θέλουμε να υπάρξει εφαρμογή των αρχών αυτών και στον τρόπο με τον οποίο το Ιερεβάν και το Μπακού αντιμετωπίζουν το θέμα και γι' αυτό οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες επηρεάζουν, θα έλεγα, αρκετά τις θέσεις τους. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ όλους. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμο σε όλες αυτές οι παρεμβάσεις. Για πέντε λεπτά διακόπτουμε για να περάσουμε στο επόμενο θέμα με λίγα λεπτά καθυστέρηση. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Βότσον, αλλά δεν μπορέσαμε να πάμε πιο γρήγορα.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 che ministro dear colleague please sit down we have to start the second point of our agenda today please Παρακαλώ, συνάδελφοι, καθίστε. Έχουμε ένα δεύτερο σημείο. Συνάδελφοι, καθίστε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, πρέπει να σας ενημερώσω ότι αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και δεν άκουσα αντιρρήσεις, θερούνται δεκτά τα πρακτικά της 9ης Μαΐου. Ξέχασα να το κάνω στην αρχή της συνεδρίασης, συγγνώμη. Έχουμε επίσης στην ημερήσια διάταξη την συζήτηση για τη σύσταση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Λάιτσκα, ο οποίος ε, είναι υπεύθυνο του τμήματος ε, που ασχολείται με την Κεντρική Ασία και τέος διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να μας ενημερώσει για τις συναντήσεις αυτές. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή μας παρακολουθεί προσεκτικά αυτές τις διαπραγματεύσεις. ξεκίνησα στις 10 Ιανουαρίου του 2010 και μας δίνει την δυνατότητα να καταθέσουμε τις συστάσεις μας, τις προτάσεις μας για τις κατευθυντήριες γραμμές ε, της ανάπτυξης των σχέσεών μας με την Μολδαβία και όποιες άλλες, σε μπάση περιπτώσει, ε, λεπτομέρειες μπορεί να περιλαμβάνει η συμφωνία αυτή. Ε, σήμερα και αύριο συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας. Έχουμε ανάμεσά μας τα μέλη της Κοινοβουλευτικής αυτής Επιτροπής οι οποίοι διέκοψαν την εργασία τους για να είναι μαζί μας. Τους ευχαριστώ για την ευγενική τους αυτή κίνηση είναι μαζί μας λοιπόν και παρακολουθούν τη συζήτηση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο αμέσως στον κύριο Γκράχαμ Βότσον, ο οποίος ε, μόλις εχρήστη από την αυτού μεγαλειότητα Ελισάβε την δεύτερη υπό της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Είναι θα έλεγα κάτι το τιμητικό, τον ευχαριστώ γι' αυτό Ζηλεύω γιατί θα πρέπει να, τον απευθύνουμε, να του απευθύνουμε το λόγο ως Sir Watson πλέον από εδώ και πέρα. Εγώ ζηλεύω γιατί δεν μπορώ να κάνω το ίδιο, δεν είμαι Βρετανός. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία των συναδέλφων από τη Μολδαβία υπό την ε, Προεδρία της ε, Κορίνα Φούσο. Μαζί με τους άλλους συναδέλφους. Θα ήθελα να χαιρετήσω επίσης τον τρόπο που διεξήχθησαν οι πρόσφατες εκλογές στη Μολδαβία, οι οποίες ε, φαίνεται ότι εκπλήρωναν ε, τα, τις διεθνείς ε, προδιαγραφές. Βεβαίως υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει, να, θα πρέπει να επιληθούν όσον αφορά την εκλογική διαδικασία, αλλά ασφαλώς ελπίζω ότι θα υπάρξει μια συνένεση όσον αφορά μια σωστή συμπεριφορά ε, στο δεύτερο γύρο των εκλογών που θα γίνουν στις 19 Ιουνίου. Παρουσιάζοντας την έκθεσή μου, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις από τις άλλες πολιτικές ομάδες, καθώς ε, και την Επιτροπή για τη συνδρομή της για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Πολλοί από εσά γνωρίζουν τη Μολδαβία πολύ καλύτερα από μένα. Η έκθεση είναι μια σύσταση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σύνδεσης. Εγώ ήλπισα, κύριε Πρόεδρε, να είμαι σε θέση να παρουσιάσω μια σύντομη έκθεση, αλλά δεν είναι τόσο σύντομη όσο έλπισα. Ε, όσο περισσότερο εγκύπτει κανείς σε τέτοια θέματα, τόσο περισσότερα πράγματα κανείς σκέφτεται ότι πρέπει να προσθέσει στην έκθεσή του. Αλλά ελπίζω ότι κάλυψα όλα τα σημαντικά θέματα και ιδιαίτερος ελπίζω ότι κάλυψα τα βασικά θέματα. Το σχέδιο του κειμένου μου, κύριε Πρόεδρε, για να το προσχέσω εν συντομία, έχει ως εξής. Τοποθετεί το, τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο μιας προοπτικής προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μακροπρόθεσμα για τη Μολδαβία και καλεί όλες τις πλευρές να σεβαστούν την ε, τιμιγορία του εκλογικού σώματος, όσο και δύσκολο, δύσκολο να είναι. Ο Τοκβίλ, νομίζω, είπε ότι ακόμα και οι ψηφοφόροι μπορεί κάποτε να τυφλωθούν, αλλά μια δημοκρατία δεν έχει την ανομιμότητα να τους το πει. Λοιπόν, η έκθεση ζητεί να υπάρξουν επαρκή πόροι εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθηθεί η Μολδαβία ούτε ώστε να επιτύχει μια συμφωνία για μια ε, εις και περιεκτική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και να προετοιμαστεί για την απελευθέρωση της ε, βίζας ε, στην προσαρμογή των οικονομικών δομών στα ε, ε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η έκθεση αναφέρει τις προδιαγραφές που αναμένουμε να εκπληρώσει η Μολδαβία και τις αναθεωρήσεις που αναμένουμε, τις μεταρρυθμίσεις που αναμένουμε. Και αναφέρεται επίσης τη σημασία της συμμετοχής των μη κυβερνητικών οργανισμών σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή στην ε, οικοδόμηση μιας πλήρως δημοκρατικής κοινωνίας. Τέλος, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει πλήρως σε αυτή τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και ιδιαίτερως ε, χαιρετίζουμε την ευκαιρία που δίνεται αυτές τις μέρες και ελπίζουμε και μελλοντικά να συζητήσουμε με μέλη του Κοινοβουλίου της Μολδαβίας για να δούμε πώς εκείνοι αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Λάβαμε κύριε Πρόεδρε μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και θα πρέπει να πω ότι ε, θα ήθελα να συστήσω στους συναδέλφους να υιοθετήσουμε τις προτάσεις ε, στο, για να τις συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Αλλά επίσης χαιρετίζω και τις υποδείξεις από τους συναδέλφους ε, που έγιναν στο σχέδιο που θα γίνουν συγγνώμη σε σχέση με το σχέδιο έκθεση που θα σας υποβάλω σήμερα. Ευχαριστώ, Σερ θα δώσω το λόγο στην κυρία Μακοβέη, συμπρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Μολδαβία. Κυρία Μακοβέη. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και επίσης, Λέμε σε ευχαριστούμε για αυτήν την τόσο πλήρη έκθεση να χαιρετήσουμε και τους έξι συναδέλφους του Μολδαβικού Κοινοβουλίου που βρίσκονται στην αίθουσα. Αποφάσισαν να έρθουν στην συνεδρίαση της ΑΦΕΤ που αφορά την συζήτηση της ε, προόδου, της προσέγγισης της ε, Μολδαβίας ε, στην Ευρώπη. Με χαρά μας να ανταλλάξουμε απόψεις εδώ στην ΕΦΕΤ. Να σας πω πάντως αμέσως ότι είμαστε στο πλευρό των αρχών της χώρας για συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά την κατάργηση της θεώρησης διαβατηρίου. Επίσης πρέπει να σας πω ότι το κλειδί είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας κάτι που είναι δύσκολο να το πετύχει κανείς. Και για αυτό τους είπαμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν προς η υλοποίηση της νομοθεσίας και όπως σας γνωρίζω από εκεί, από την περιοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι και αυτό είναι η μεγάλη δοκιμασία. Πάντως θεωρούμε ότι χρειάζεται και η οικονομική υποστήριξη αυτή η προσπάθεια. Επίσης έχω να σας πω ότι η εφαρμογή πάει να πει η φάση κατά την οποία ο κόσμος βλέπει τη διαφορά στη χώρα επί τόπου. Οπότε να σας πω πως είναι επίση πάρα πολύ σοβαρό το να ζυγίζουμε το τι έχει καταφέρει η χώρα μέχρι τώρα, γιατί μέχρι τώρα τα έχει πολύ καλά καταφέρει. Να είναι η ανατολική εταιρική σχέση και εμεί επομένω ω εταίρου που βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς, να ζυγίζουμε, να υπολογίζουμε τα όσα πετύχανε και οπότε βεβαίως και αυτοί έχουν λάβει τις ευθύνες τους και βεβαίως έτσι θα πρέπει να κρυθεί και η συνέχεια τώρα όσον αφορά τα περαιτέρω εμπόδια εμείς στηρίζουμε αυτή τη χώρα ή στις προσπάθειες να υπερκειάσουν τα προβλήματα και επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την υπερδυνστερία. Θα γίνει πάρα πολύ σύντομα μια σχετική συνάντηση. Και αυτό πρόκειται να μας οδηγήσει σε ένα βήμα προόδου προς την επίτευξη των στόχων προσεγγίσει στην Ευρώπη και βεβαίω είναι πάρα πολύ καλό το ότι υπάρχουν αυτές οι επίσημες επαφές που ήταν κάτι που δεν γινόταν στο παρελθόν. Είναι επομένως πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα έχουμε διεθνή αστυνομική δύναμη γιατί από το 1992 και μετά δεν είναι καμία προστριβή, σύγκρουση, λέμε για παγωμένες συγκρούσεις. Για να δούμε, περί τίνος πρόκειται πραγματικά. Ίσως τα πράγματα δεν είναι τόσο συγκρουσιακά και ίσως θα πρέπει και οι πολιτικές αποφάσεις να αντικατοπτρίζουν την κατάσταση. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μακοβέη. Συμφωνείτε λοιπόν και συμφωνώ και εγώ με τον κύριο Λάιτσα και να κερδίσουμε λίγο χρόνο η παρέμβασή σας θα ακολουθήσει τις παρεμβάσεις των άλλων συναδέλφων και θα είναι και ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις και απάντηση στις ερωτήσεις σας. Δίνω το λόγο λοιπόν αμέσως στον κύριο Πρέντα, ο οποίος εκπροσωπεί τον κύριο Ουν, Ουνγκουρεάνου, που είναι σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω τους συναδέλφους ε, βουλευτές της ε, Μολδαβικής Δημοκρατίας που είναι ανάμεσά μας σήμερα. Θα ήθελα να πάρω το λόγο εξ ονόματος του κυρίου Ουγγουρεάνου που είναι σκιώδης εισηγητής της ομάδας μας για την έκθεση αυτή. Ο συνάδελφος προσπάθησε και καταλήξαμε σε μια κάποια συμφωνία. Ο κύριος Γκουρεάνο θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την πρόταση στην οποία κατέληξε. Στο κείμενο ξαναβρίσκει κανείς τα βασικά στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν στις ε, συζητήσεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει μέχρι τώρα ανάμεσα στον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή. Ο κύριος Σαγκουρεάνο θεωρεί ότι η Μολδαβική Δημοκρατία θα πρέπει να στηριχθεί στις διαδικασίες τις οποίες έχει αναλάβει έτσι ώστε κάποια μέρα να μπορέσει να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελε όμως ο κύριος Σουγκουρεάνο να κάνει τρεις ίσονες παρατηρήσεις που εκπροσωπούν και το σύνολο της ομάδας μας. Καταρχάς σχετικά με το 1C αγγλικό. Εκεί γίνεται αναφορά στην σχέση με τις γειτονικές χώρες. Θεωρεί ο κ. ότι πρέπει να υπάρξει αναδιατύπωση και θα καταθέσει μια τροπολογία προς την κατεύθυνση αυτή σχετικά με το 1G αγγλικό. Εκεί που γίνεται αναφορά στην υπερδνηστερία σαν αναπόσπαστο τμήμα του εδάφους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και μία τελική παρατήρηση σχετικά με την πολιτική στον τομέα της έρευνας. Το ένα Q αγγλικό. Θεωρεί ο κύριος Σουγκουρεάνου ότι στα πλαίσια αυτού του εδαφίου θα πρέπει να υπάρξει αναφορά σε μια ευρύτερη προβληματική της ενεργειακής πολιτικής και στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τροφοδοτείται σε ενέργεια και γι' αυτό θα καταθέσει τις αντίστοιχες τροπολογίες για τα τρία αυτά σημεία. Εποφελούμε, μιας και έχω το λόγο, για να μιλήσω τώρα ε, προσωπικά και όχι εκ μέρους του κυρίου Ογκουρεάνου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βότσον και θα ήθελα να εκφράσω και την ικανοποίησή μου για, τις, ε, για τη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών στη Μολδαβική Δημοκρατία. Θα ήθελα επίσης όλα να καταλήξουν στις ε, επιθυμητές ε, γενικά συνθήκες και σχετικά με το θέμα της υπερνηστερίας τους τελευταίους μήνες πήραμε ορισμένα ενθαρρυντικά μηνύματα θα έλεγα από την υπερνηστερία. Πρόκειται για μια σύγκρουση η οποία βρίσκεται στις θύρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζουμε από ε, πολύ σύντομα να βελτιωθούν τα πράγματα, να υπάρξουν πιέσεις. Ξέρουμε ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες επαφές ανεπίσημες και από ό,τι φαίνεται οι επαφές αυτές ε, αρχίζουν να αποδίδουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η σύγκρουση αυτή να αποτελέσει παρελθόν το θέμα της υπερδνηστερίας δηλαδή. Να υπογραμμίσω επίσης και κάτι το οποίο έχει ήδη πει η κυρία Μακοβέη σχετικά με το πρώτο εδάφιο λέγεται ότι η Μολδαβική Δημοκρατία έχει την δυνατότητα να είναι ένα υπόδειγμα επιτυχίας στην περιοχή γειτονίας. Και θέλει συνάδελφος Μακοβέη να πούμε ότι η Μολδαβία είναι ήδη ένα success story. Όχι ότι θα γίνει κάποτε. Λοιπόν, πράγματι αυτό μπορούμε να το αναδιατυπώσουμε. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε χρόνια για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. <coughs> Αυτό το κάνουμε ήδη με την Τουρκία και ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Κύριος Πάσκου, δεύτερος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και σκιώδης εισηγητής για τη Σοσιαλιστική Ομάδα Πάσκου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τον Σερ Γκρέαμ Βότσον. Μια αυτό το ε, σχέδιο εκθέσεως καλύπτει όλα όσα συζητήσαμε όπως ε, αναγνώρισε και ο κύριος Πρέντα διότι κατά τη γνώμη μου πρόκειται για μια έκθεση που θα συμβάλλει πάρα πολύ σημαντικά ε, αυτή την κρίσιμη στιγμή που πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με όλα αυτά τα προβλήματα που αναδύονται στην περιφέρεια της Ευρώπης και άρα θα πρέπει να επαγρυπνούμε όσον αφορά το τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε με αυτές τις χώρες όπως τη Μολδαβία γιατί θα πρέπει με τις αποφάσεις μας να μην εγκαταλείπουμε την ξεχασμένη Ευρώπη ε, όσο και αν είναι πια λίγε αυτέ που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, όπω η Μολδαβία και τώρα για να δούμε όσον αφορά αυτό το σχέδιο τη έκθεση, όπω σήμερα έχει το κείμενο το οποίο νομίζω ότι θίγει τι βασικέ πτυχέ του θέματο, τα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Μολδαβία. Θεωρώ ότι με αυτή την έκθεση μπορούμε να ε, ελκύσουμε την προσοχή της ε, χώρας για να προσέξει το τι γίνεται. Ε, μια που πρόκειται για ιστορική στιγμή για τη χώρα και επομένω, μια που είναι τόσο σημαντικέ ε, οι ώρε, θα πρέπει και εκεί να καταβληθούν προσπάθειε ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από την ευκαιρία που του προσφέρει η ιστορία. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για την υποψηφιότητα. Θα πρέπει οι ίδιοι οι Μολδαβοί να δώσουν απαντήσεις εις όλα όσα απαιτούνται. Κατά γνώμη μου, όλα αυτά τα λέει το κείμενο πάρα πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Και επίση, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι θα βοηθήσω όσο μπορώ τον συγκητή, ω σκιώδη που είμαι εγώ, επίση και η πολιτική μου ομάδα γενικότερα ενδιαφέρεται να καταλήξουμε σε μια αξιόλογη έκθεση για την υποσχέτα αυτή τη ε, χώρα που μόνο θετικά έχει να δώσει. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχει το λόγο ο κύριο Σούλτς, Σκιώδη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους από τη Μολδαβία και θα ήθελα να πω ότι η έκθεση που υπέβαλε ο κύριος Βόκτσον είναι πραγματικά πολύ περιεκτική και ισορροπημένη και μόνο σε λιγοστά σημεία χρήζει κάποιων διευκρινήσεων ή συμπληρώσεων. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό και αυτό το δείχνει η έκθεση η δημοκρατία της ε, Μολδαβίας ε, μεταξύ των έξι χωρών που έχουμε στην Ανατολική Γειτονία δείχνει ένα ξεκάθαρο προσανατολισμό προς την Ευρώπη και έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες. Γι' αυτό ξεχωρίζει μεταξύ αυτών των χωρών, εάν τη συγκρίνουμε με, τα, με τις άλλες χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Στην ίδια την έκθεση θα πρέπει να γίνει μια επισήμανση ε, στη στρατηγική ε, της ε, Μαύρης Θάλασσας και νομίζω ότι είναι σημαντικό σε σχέση με την υπερδνηστερία και με τις διαπραγματεύσεις 5 συν 2. Δηλαδή ότι απαιτούμε η Ρωσία στην περίπτωση αυτή να έχει ένα πιο ενεργό και επικοδομητικό ρόλο. Γιατί μέχρι στιγμής ε, δεν εφαρμόστηκαν δηλώσεις του Πρόεδρου Μετβέντεφ. Ε, σε σχέση με τη Βίζα, λέχθηκε ότι ε, σταμάτησε η έκδοση των ε, διαβατηρίων ε, και θεωρώ ότι αυτό πραγματικά υπονομεύει το, τη Συμφωνία Σέγγεν. Γι' αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι δεδειγμένη μια συνολική οικονομική υποστήριξη της Μολδαβίας σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σούλτς. Τώρα... Non c'è. Allora l'onorevole Belder, relatore... Ο κύριος Χατζηγεωργίου δεν είναι εδώ, όμως ο κύριος Μπέλτερ, σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ε, και ευχαριστώ μάλλον που μου επιτρέψατε να θέσω μία ερώτηση. Ε, νομίζω ότι η έκθεση του κ. Βότσον είναι πραγματικά καλή. Στις, ε, πιστεύω ότι πραγματικά σας αξίζει ο τίτλος που σας απονεμήθηκε, ο τίτλος τιμής. Τώρα, συγχαρητήρια. Ε, πριν από λίγο καιρό έμαθα ότι υπάρχει ένα λεγόμενο non-paper και την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε για το ζήτημα της υπερδυνιστερίας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή αλλά και τον κύριο Λάιτσεκ ε, ε, τι σημασία προσδίδεται σε αυτό το non-paper γιατί οι διάφορες αναλύσεις που έγιναν εκφράζουν κάποιες ανησυχίες και θεωρείται ότι είναι προβληματική κατάσταση αν δούμε τι γίνεται στην ε, Ρωσία. Και ίσως ε, με τον τρόπο αυτό απειλείται ο ευρωπαϊκός ε, δρόμος της Μολδαβίας. Δεν αναφέρεται τέτοιο στο κείμενο του κυρίου Βότσον, αλλά θα ήθελα ο κύριος Λάιντζεκ να μας πει πώς αντιμετωπίζει το γερμανικό non-paper. Πρόκειται για ένα γερμανικό κείμενο, όχι ένα ευρωπαϊκό κείμενο αλλά ωστόσο είναι σημαντικό στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 5 συν 2. Γιατί υπάρχουν ορισμένα θέματα, όπως για παράδειγμα η απόσταση των στρατευμάτων από την υπερνηστερία. Και ε, τα θέματα αυτά δεν τίθενται εδώ. Ε, νομίζω ότι αυτό το Noin Paper θα μπορούσε να ασκήσει μεγάλη επιρροή και η ρωσική θέση ίσως μπορεί να σκληρινθεί εις βάθος προηγούμενων συμφωνιών που προβλέπουν μια αποστρατικοποίηση της ε, περιοχής. Ένα σημαντικό τμήμα των σχέσεων μεταξύ Μολδαβίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι διαπραγματεύσει για τη Βίζα. Ε, πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, ε, τι γίνεται με την προσαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων. Ορισμένες ε, ρήτρε ε, θεωρώ ότι είναι υπερβολικές όσον αφορά τις ε, διακρίσεις κατά του θρησκεύματος. Αλλά αν περιμένουμε ότι περιμένουμε πραγματικά η σχετική νομοθεσία στη Μολδαβία να πάει πιο μακριά από την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά για παράδειγμα τις διακρίσεις. Κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συζητούσαμε στην Επιτροπή Διακοινοβουλευτικής Συνεργασίας την κατάσταση στη Μολδαβική Δημοκρατία και συμφωνήσαμε ότι και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα βρισκόμαστε λόγω της οικονομικής κρίσης σε μια δύσκολη φάση. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι για τη Μολδαβία υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κάποια ευκαιρία γιατί τα τρία θεσμικά όργανα αντιμετωπίζουν το θέμα με σοβαρότητα το Συμβούλιο στο νέο έγγραφό του είναι ιδιαίτερα σοβαρό θα έλεγα στην υποστήριξη που δίνει σε αυτούς που έχουν κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο. Έχουμε μιλήσει για την αιρεσιμότητα αρκετές φορές στο παρελθόν. Μετά από την Ουγγρική Προεδρία νομίζω ότι και η Πολωνική θα το αντιμετωπίσει το θέμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο κύριος Βότσον προετοίμασε μια εξαιρετική έκθεση. Το μόνο που θα ήθελα να πω εδώ είναι ότι μιλάμε συνεχώς για την δυνατότητα δράσης ε, από κοινού με τις γειτονικές χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο αναλυτικοί, σημειώνοντας την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Έχει υπάρξει πρόοδος. Ζητούσαμε πολλά τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχε συμβεί κάτι σημαντικό, τώρα όμως έχουμε κάποια ξεκάθαρα μηνύματα για τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δυνατότητα που έδωσε να προχωρήσουν τα πράγματα. Για τον κύριο Λάπτσακ. Δεν γνωρίζουν πολύ ότι η Μολδαβία είναι υψηλά στην πολωνική ατζέντα που είναι η προεδρία που θα ακολουθήσει. Διαρωτώμεθα λοιπόν για το τι αποτελέσματα μπορούμε, σε τι αποτελέσματα μπορούμε να καταλήξουμε κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας αυτής. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω εσάς, γνωρίζετε την περιοχή κύριε Λάιπτσακ, τι πιστεύετε εσείς ότι είναι το αποτέλεσμα στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε το πιο σημαντικό. Πείτε μας δύο-τρία πράγματα στα οποία πρέπει να καταλήξουμε τους επόμενους έξι μήνες για να πούμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Πείτε μας λοιπόν ποια είναι ποιοι είναι οι στόχοι αναφοράς τους οποίους θα πρέπει να επιδιώξουμε να πετύχουμε σαν επόμενη Προεδρία. Ευχαριστώ κύριε Ταυσκόφσκι. Η κυρία Φούζου, συμπρόεδρος της Αντιπροσωπείας με τη Μολδαβική Δημοκρατία. Φούζου. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει η κυρία Φούζου. Εκ μέρους της ε, αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου μας χαιρετίζουμε την έκθεση της ΑΦΕΤ και ευχαριστούμε τον κύριο Βότσον για το έργο το οποίο επετέλεσε. Έχουμε να σας δηλώσουμε τα εξής. Θεωρούμε πως οι θέσεις που εκφράζει η έκθεση είναι ορθές και αποτελεσματικές για την επίτευξη των στόχων μας. Ο διάλογος όλων των πολιτικών κομμάτων είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, μας απασχολεί, όπως αυτό ανέκαθεν ίσχυε. Αυτό άλλωστε αναφέρεται και στο σύνταγμά μας και το αναφέρει και ο κύριος Βότσον. Όσον αφορά τώρα τις ε, πρόορες εκλογές Θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστικό. Μόλις δύο χρόνια έχουν, έχει, διανύσει αυτό το κοινοβούλιο. Πάντοτε η κυβέρνηση έχει επαφές με την αντιπολίτευση και βρισκόμαστε σε διάλογο. Όμως προσπάθειες συμβασμού και συνένεσης ε, δεν έχουν πιάσει τόπο, οπότε ε, ξέρετε ότι έχει επιληφθεί το συνταγματικό δικαστήριο ούτως ώστε να επιληφθεί ένα θέμα συνταγματικής ε, τάξης που έχει ε, αναδειθεί στην χώρα. Ε, αυτό το θέμα δεν μας κολακεύει, οπότε το συνταγματικό δικαστήριο πρόκειται να γνωμοδοτήσει λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις τις προτάσεις τα όσα έχουν να προτείνουν ε, ας πούμε και η Επιτροπή της ε, Βενετίας. Οι διαμετεύσεις πέντε συν έχουμε τώρα το στιγμή Έτσι μπορούμε να, θεωρήσουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε όσον αφορά για την επίλυση της προστριβή για την υπερτινιστερία. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιτευχθεί πιο έντονα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι θεωρίε διαβατήριων. Ε, Επίση θεωρούμε ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσει για τη ζώνη ευθύνων συναλλαγών και όσον αφορά τώρα το στόχο στην επίτευξη της προσέγγισης στην Ευρώπη και αυτό είναι μια προτεραιότητα για μας. Ε, επιθυμούμε να ενθαρρυνθεί η κινητικό της επίσης, να έχουμε νόμιμη μετανάστευση και ελεγχόμενη μετανάστευση. Και επομένω κατά τον τρόπο να μπορέσουμε να τονώσουμε τις εμπορικές μας συναλλαγές όσον αφορά τώρα ε, τις προτεραιότητες μας για την περίοδο 2011 2014 εδώ έχουμε θέσει μια σειρά στόχων ο κοινό στόχος ξέρουμε ότι υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη επαγγελματική δικαιοσύνη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα Επίσης ε, έχουμε εγκρίνει ένα νομοθετικό πρόγραμμα έτσι θα πληρούμε περισσότερο τα κριτήρια τα οποία θα μας δώσουν ευκαιρία να ωφεληθούμε από την κατεύθυνση της βίζας Επίσης το Κοινοβούλιο της χώρας θα προχωρήσει σε μια σειρά έγκρισης νόμων που θα αφορούν ακριβώς την προσέγγιση στην Ευρώπη Υπήρχε ένα πρόβλημα με το νομοσχέδιο ε, για τι μηνύες διακρίσεις, γιατί θέλουμε να είναι ανοιχτική η κοινωνία μας, αλλά υπήρχε ένα προβληματάκι και δεν θα επιληθεί. Και εκτός από τη δημόσια προβληματική θα υπάρξει και για το πρόγραμμα TAEX ένα σεμινάριο το οποίο θα οργανωθεί και αφορά ακριβώ την αποφυγή δυσμένων διακρίσεων. Ε, επίσης, Έχουμε τις ε, προτεραιότητες του Υπουργείου Μεταφορών για να μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη κινητικότητα. Να διευκολύνουμε δηλαδή τις ε, μετακινήσεις και των δικών μας ε, υπηκών αλλά και τις, τους Ευρωπαίους που θέλουν να έρθουν. Μας βοηθούν οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει ανοιχτός διάλογος Επίσης ε, υπάρχει και η ενημερωτική εκστρατεία για να ξέρει ο κόσμος τι πάει να πει η Συμφωνία Σύνδεσης. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να στηρίζει τις μας ο λαός. Ούτως ώστε όλοι μαζί να πετύχουν τελικό στόχο που είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ε, εγγυόμαστε εμείς το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας σήμερα, σήμερα περισσότερο από ποτέ η συμμαχία για την ευρωπαϊκή ένταξη που κατέχει την εξουσία θέλει να τηρηθούν όλες μας οι δεσμεύσεις, να κάνουμε ό,τι μεταρρυθμίσει χρειάζεται, τόσο ώστε η χώρα και οι πολίτες να μπορούν κάποια στιγμή να ζήσουν σε μια χώρα που είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπορούμε να ζήσουμε με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το εμπορικό κινητικό δίκαιο και νομίζουμε ότι ο δρόμος που μπροστά μας δεν είναι πάρα πολύ μακρύς, οπότε και γι' αυτό και ε, θα προχωρήσουμε χέρι-χέρι με την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την περίπτωση. Eh, eh, Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Λάιτσακ που θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις και θα απαντήσει ταυτόχρονα τις ερωτήσεις που του υπευλήθησαν. Παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και πάλι καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ όχι μόνο υπό την ιδιότητά μου ως Managing Director της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, αλλά ως βασικός διαπραγματευτής της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Μολδαβίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να ξεπίσω αυτή την ευκαιρία για να σας δώσω πρώτες αντιδράσεις για το σχέδιο έκθεσης που προετοίμασε ο κύριος Βότσον και για να απαντήσω ενδεχομένω στις ερωτήσεις σας που αφορούν την ε, κατάσταση, το επίπεδο της συμφωνία ε, ε, Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας. Θα ήθελα να χαιρετήσω το ενδιαφέρον που έδειξαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Συμφωνία και την πορεία διαπραγματεύσεων. Στην αρχή Τη σύσταση αναφέρεστε στη δυνατότητα της Μολδαβίας να γίνει το success story της Ευρωπαϊκή πολιτικής γειτονία. Και πράγματι θα ήθελα να επικυρώσω ότι οι διαπραγματεύσεις ε, εξελίχθηκαν πολύ ήπια από το 2010. Υπήρξαν έξι γύροι διαπραγματεύσεων στο Κισινάου και στις Βρυξέλλες Αλλάξ, και η συνεργασία με την ομάδα της Μολδαβίας ήταν εξαιρετικά καλή. Στις 5 Ιουλίου θα υπάρξει ο επόμενος γύρος στις Βρυξέλλες και με την Ατάλια Γκέρμαν, υφυπουργό ε, συντάξαμε την αναφορά η οποία υπευλήθη στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας το Μάιο. Επίσης ε, ε, διανύμαμε αυτή την έκθεση για την, σε εσά για τη σημερινή συζήτηση. Πριν αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία που αναφέρονται στο σχέδιο σύστασης, θα πω ότι καλύψαμε Πολλού τομεί συνεργασία, αμοιβαία ενδιαφέροντο. δηλαδή την πραγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πραγωγή των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, συνεργασία στον αγώνα κατά των διακρίσεων, κατά πολέμηση τη διαφθορά, ε, ενεργειακή συνεργασία κλπ. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω ορισμένα θέματα, συγκεκριμένα θέματα των συστάσεων. Πρώτον, αναφορά στη μακροπρόθεσμη ε, προσχώρηση της Μολδαβίας. Η Μολδαβία προσδίδει μεγάλη σημασία στην ευρωπαϊκή τη ταυτότητα και οι συμφωνίες λένε στο προήμιο ότι οι ευρωπαϊκές ε, φιλοδοξίες της, ε, δρώνονται στο λαό της ε, Μολδαβίας και αυτό καθορίζει, θεωρώ, τις μελλοντικέ εξελίξεις και μπορεί να γίνει αποδεκτό από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Θα σημειώσετε στην πρόσφατη ανακοίνωση ε, αναφερθήκαμε ξεκάθαρα στις αξίες στις οποίες έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι οι ίδιες αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της συνθήκης, στο, άρθρο 8, στο οποίο βασίζεται το άρθρο 8 και το άρθρο 49. Μαζί με τις άλλες χώρες μέλη θα ε, προσπαθήσουμε να καλύψουμε τόσο τις ε, φιλοδοξίες της Μολδαβίας όσο και την προσφορά εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά δηλώσαμε την προθυμία μας να δώσουμε περισσότερα σε χώρες που έκαναν, που έπραξαν πολλά. Ε, ε, η Μολδαβία έδειξε μεγάλη βούληση για να προβεί σε μεταρρυθμίσεις και ε, έγινε και θα ήθελα να τονίσω ότι πράγματι η δημοκρατία της Μολδαβίας έχει το δυναμικό να είναι ε, ε, μια χώρα που θα βερθεί από τη νέα αυτή προσέγγιση γιατί πραγματικά έδειξε υψηλό επίπεδο δέσμευσης για να τηρήσει τις ε, προδιαγραφές της οικονομικής ολοκλήρωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το θετικά σε αυτή την πολύ θετική στάση της Μολδαβίας. Επίσης αναφέρεστε στο κείμενό σας στην επίλυση του, της σύγκρουσης υπέρ της Και είμαι ευτυχής που μπορώ να σας πω ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου της Ολομέλειας στο Κισινάου αριστικοποίησαμε το κείμενο για τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία εν σχέση με την ΚΕΠΑ, η οποία περιλαμβάνει ένα άρθρο, το οποίο περιλαμβάνει ένα άρθρο για την περιφερειακή σταθερότητα και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 5 συν 2 ε, και την υπερνηστερία μπορώ να επικυρώσω ότι εργαζόμαστε σκληρά για να περάσουμε στην επόμενη φάση, δηλαδή την ανάληψη επίσημων συνομιλιών που έχουν σαν στόχο την πολιτική διαθέτηση του ζητήματος της τρανσμυστερίας ε, που θα ενθαρρύνει μια νέα φάση μετά από πέντε έτη διακοπής των συνομιλιών. Ο επόμενος γύρος του των συνομιλιών του 5 συν 2 σχεδιάζεται για την προσεχή εβδομάδα, την Τρίτη στη Μόσχα και θα πάμε εκεί με την φιλοδοξία να εξαγγείλουμε την ανάληψη των επίσημων συνομιλιών που είναι τέλος σημαντικό για τη Μολδαβία. Τώρα όσον αφορά το διάλογο για τη Βίζα που είναι σημαντικό στοιχείο που αναφέρεται στην, στο κείμενο και την απελευθέρωση από την υποχρέωση των θεωρήσεων. Θα ήθελα να πω το κείμενο προβλέπει σημαντικέ διατάξει σε σχέση με το διάλογο για τη Βίζα και μαζί με την ομάδα διαπραγμάτευση για τη Μολδαβία αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις σε σχέση με αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή οι συζητήσει έχουν προχωρήσει το κείμενο αυτό θα διατυπωθεί υπό το πρίσμα αυτών των συζητήσεων όσον αφορά τις ε, προϋποθέσεις μιας ελεύθερης ε, μετακίνησης των, πολιτών της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έγινε αναφορά στην νομοθεσία κατάργησης των διακρίσεων και πράγματι αυτό είναι ένα τμήμα της συζήτησης που σχετίζεται με την απελευθέρωση από την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίων ε, και, αλλά ε, το Κοινοβούλιο απέσυρε το σχέδιο πρόταση το Μάιο. Παρόλα αυτά ε, μας είπαν ότι το σχέδιο νόμου θα επαναυποβληθεί προς έγκριση στο Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του χρόνου και αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Ε, βρισκόμαστε λοιπόν σε μια προχωρημένη φάση όσον αφορά τη βίζα το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υποβληθεί από τον Επίτροπο Μάλστρομ τον Ιανουάριο και αναπόκειται στην κυβέρνηση της Μολδαβίας να εφαρμόσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις με ένα περιεκτικό τρόπο, ούτω ώστε οι χώρες μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν για την άρση των υποχρεώσεων θεώρησης διαβατηρίων για τη Μολδαβία. Φυσικά δεν είναι δυνατό να προβλέψουμε την καταληκτική ημερομηνία για αυτή τη διαδικασία, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι στα θέματα αυτά η ποιότητα είναι πολύ περισσότερο σημαντική από την ταχύτητα. Τώρα, όσον αφορά το DCFTA, γνωρίζουμε και θα ήθελα να πω ότι η κυβέρνηση της ε, Μολδαβίας θέλει να ξεκινήσει τις ε, διαπραγματεύσεις το ταχύτερο δυνατό. Ε, δηλαδή πρόκειται για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που να είναι περιεκτική και να πηγαίνει εις Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συνεργάζεται με την Κομισιόν προς αυτό το στόχο και έχουν υποβληθεί συστάσεις κλειδί το φθινόπωρο ούτως ώστε να αρχίσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις για τη ζώνη ελεύθερου εμπορίου και τώρα η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει αυτές τις συστάσεις και προετοιμάζεται μια διαπραγματευτική εντολή η οποία έχει υποβληθεί την Άνοιξη στο Συμβούλιο και οι ιστορικές διαδικασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί άρα περιμένουμε προ την τελική έγκριση. Επίσης γίνεται αναφορά στο πρωτόκολλο για τη συνεργασία και τη συμμετοχή της Μολδαβίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ε, στις ευρωπαϊκές θεσμικές υπηρεσίες. Εδώ ε, γίνονται κάποιες συζητήσεις και εν ώψη της προσεχούς ολομέλειας η ομάδα θα συντάξει ένα κεφάλαιο το οποίο θα αναφέρεται στη συμμετοχή της Μολδαβίας στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, προέρχεται στην κατάθεσή της. Επίσης γίνεται αναφορά στη συνέχεια της καλής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και στη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε όσον αφορά τις θεσμικές διατάξεις της συμφωνίας και θα συμπεριλάβουν την διατύπωση που αφορά την κοινοβουλευτική διάσταση. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίσουν ε, και γίνεται επίσης ε, ε, μνήμα ε, στην ε, ενημέρωση των Ευρωπαίων Βουλευτών και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση της Επιτροπής ΑΦΕΤ ε, ή προς τους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης βρίσκει συνεχή επαφή με τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. τελευταία ερώτηση, δύο ερωτήσεις που τέθηκαν στις συζητήσεις σχετικά με το γερμανικό non-paper όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία ε, κάπως ε, ε, αχώδη περίοδο προετοιμασίας της συνάντησης της Μόσχας. Πολλά κείμενα παρασκευάζονται και παρουσιάστηκε ένα κείμενο, ένα paper που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση της Μολδαβίας, της Ρωσίας, την Ουκρανία, τον ΟΑΣΕ και επίσης υπάρχει ένα non-paper το οποίο διατυπώθηκε, εκπονήθηκε στο Βερολίνο, βεβαίω το είδα και θεωρώ ότι θα γραμμίζεται με τις γενικές γραμμές ε, της πολιτικής, επίλυσης, ε, πολιτικής λύσης για την υπερδνηστερία. Και παρόλο που η Γερμανία δεν είναι μέρος του 5 2 πλαισίου, θεωρώ ότι είναι επικοδομητική εισφορά της. Τέλος, όσον αφορά τα αποτελέσματα ε, κατά τη διάρκεια της Πολωνικής ε, Προεδρίας, ε, έχουμε επίγνωση της σημασίας που προσδίδει η Πολωνική Προεδρία στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ καλά και εν γέννη όσον αφορά την Πολωνική Προεδρία, αυτό το οποίο θα ήθελα να δω είναι μια επιτυχημένη συνάντηση κορυφής το Σεπτέμβριο της ε, Βαρσοβίας που θα δώσει ε, περαιτέρω ρεθίσματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής γειτονίας και θα δώσει αυτά αποτελέσματα ειδικά για την Μολδαβία. Ε, πρόκειται εμεί να συνεργαστούμε προς τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη ζώνη ελεύθερου εμπορίου και ε, προς την κατεύθυνση της, ε, ε, των θεωρήσεων, της απελευθέρωσης από την υποχρέωση θεώρηση των διαπατηρίων. Αυτά θα σημεία είναι ιδιαίτερως ζωτικά στο πλαίσιο του προγράμματος για την πολιτική ανατολικής γειτονίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Λάιτσακ όχι μόνο για την ενημέρωση και το briefing που προετοιμάσατε, αλλά και για τη διαθεσιμότητά σας να είσαστε ανάμεσά μας σήμερα και οπότε έχουμε να συζητήσουμε τόσο σημαντικά θέματα που είναι τμήμα και των δικών σας ευθυνών. Θα ήθελα να καλέσω τώρα τον εισηγητή, τον κύριο Βότσον, να κλείσει τη συζήτηση. Έχετε το λόγο κύριο Βότσον. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις ε, ε, ε, ιδέες που προτείνανε με κανείς ρίξει μια ματιά στο κείμενο κανείς θα βρει βέβαια ε, το ότι έχουν παρισφρήσει κάποια τεράτουργήματα τουργήματα που το συμπήρασμε στο Β' θα χρειάζεται να δούμε πώς θα έχουμε την ομαλή ροή εμπορευμάτων. Το δεν το λέει καλά, τα στα αγγλικά είναι λάθος. Ε, αυτή η λέξη που λέει trafficking αντί για traffic ε, πάνε να πήγει λαθρεμπόριο τέλο πάντων. Λαθρέα παράνομη διακίνηση. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν λέμε για την ε, Μολδαβία ότι θέλουμε να πετύχει. Έχει ήδη πετύχει στα πλαίσια τη γειτονία προ Ανατολά. σω μπορούμε να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που ε, πετυχαίνει η πολιτική μας προς Ανατολάς και θα έχουμε και στη συνέχεια επίσης πάρα πολύ θετικό είναι ότι η Πολωνική Προεδρία ενδιαφέρεται εντόνως για όλη αυτή τη διαδρομή με τον Σικόρσκι μίλησα, τον Ιπέξ και μου ξέρω και έμαθα ότι έχει δεσμευθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να προχωρήσουν τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Κυρία Μακοβέη μας μίλησε για την σύγκρουση που έχει παγώσει βεβαίως και πολλά θα παιχτούν την επόμενη εβδομάδα ή στην συνάντηση ή στην Μόσχα για το τι θα γίνει στα πλαίσια της των 5 συν 2 τώρα για αυτά που είπε Συνάδελφος Μπέλντερ, ε, έχετε δίκιο για το Μέντεβεντεφ. Να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Ίσως μπορέσουμε κάπως να συμβάλλουμε όσον αφορά το 5 2 καθώς προχωράει και η εκθεσή μας επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά τον κύριο Μπρέντερ και τον κύριο Πάσχου για τόσα επρότειναν. Και Περιμένω πώς και πώς τις ε, τροπολογίες τους, γιατί όπως και εσύ είπες πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή, πολύ κρίσιμη για τη Μολδαβία. Έχουμε και άλλα θετικά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι και θα έπρεπε εγώ να τα έχω βάλει όσον αφορά τη στατική της Μαύρης Θάλασσας, όπως το είπε ο κύριος Σούλτς, ίσως όπως ο Βασμπέλτερ είπε αλλά και άλλοι θα έπρεπε την παράγραφο μη για την πολιτική των διακρίσεων κάπως να την κάνουμε πιο δυναμική. Τη διατύπωση πιο ζωντανή για να πούμε ότι δηλαδή ενδιαφέρομαστε πώ και πώ για το να υπάρχει πρόοδο στην Μολδαβία όσον αφορά την καταπολέμηση των δεσμών διακρίσεων και επίση την κυρία Φούζου την ευχαριστώ και αυτή για τα όσα μα ανέλησε όσον αφορά το πώς έχει προχωρήσει η νομοθετική προσπάθεια για αυτό το θέμα ή στην χώρα. Ε, επίση, Πρόεδρε, όπω είπε ο κύριο Στασκόφσκι, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αναλυτικοί, πιο συγκεκριμένοι, για τις προσπαθίες της χώρας σε διαφορετικούς τομείς να προσεγγίσουν αυτά που θέλουμε. Έχουμε επίσης και την αναμονή της ε, απόφαση του Εγγοντικού Δικαστηρίου που θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη και επίσης και η κυρία Φούζου και αυτά μας τα εξήγησε. Κύριε Λάιτσακ, μάλιστα αυτό αυτά τα οποία είπατε και όπως τα είπατε όσον αφορά το ότι πρόκειται εκεί πέρα για κάτι σαν ένα εργοτάξιο ή είναι ένα εργοστάσιο πραγματικά και όπως ε, πολλοί από μας θα μπορούσαν να πούνε το ίδιο ισχύει και για την υπηρεσία τη εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκείνη είναι έτσι, και εκείνη είναι εργοτάξιο. Όμω τα εργοτάξια τα αυτά θέλουμε να υπάρξει γρήγορη πρόοδο. Άρα, συνεχίζουμε λοιπόν την πορεία μα για αυτή την εκθεσία. Ο πρόεδρο. Σερ Γκράμ, ευχαριστούμε. Έχουμε εδώ το χρονοδιάγραμμα που αφορά τι εργασίε μα, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η παρουσίαση των τροπολογιών στις 21 ε, Ιουνίου το μεσημέρι, στις 12 Ιουλίου θα γίνει η συζήτηση των τροπολογιών και θα γίνει η ψήφιση στην Επιτροπή μας που προβλέπεται να γίνει στις 13 Ιουλίου και επίση στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου θα γίνει η ψήφιση της εκθέσεως. Ευχαριστούμε όλους τους έλαβαν μέρος. Ιδίως δε τον διευθυντή, τον κύριο Λάιτσακ. Μεγάλη του καλοσύνη το ότι κάθεσε όλη αυτή την ώρα εδώ πέρα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Περνάμε τώρα για να κερδίσουμε λίγο την καθυστέρηση που έχουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη το σχετικό με τον οικονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης. Α, για μια στιγμή κάποιος έχει ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Μπροκ. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Μπροκ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω εξ ονόματος επίσης των συναδέλφων ε, Γουαλτιέρη και Νταφ γιατί είμαστε τελευταία συνάντηση Κόζακ και νομίζω ότι είναι αναγκαίο ε, να πούμε ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας σε μια σύντομη διατύπωση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και αυτό σε σχέση και με τα εθνικά κοινοβούλια και νομίζω ότι εδώ συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ε, εγκρίνουμε αυτό το κείμενο της προσεχής εβδομάδας, να ψηφίσουμε αυτό το κείμενο. Ε, δεν ξέρω ε, ίσως να πάρουμε σχετική απόφαση να διατυπωθεί το κείμενο αυτό και στη συνέχεια να το επικυρώσουμε, ίσως πριν από την Ολομέλεια. Θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Μπροκ και θα ήθελα να σας παρακαλέσω εσείς ο ίδιος να εισηγηθείτε ένα ψήφισμα για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει δεκτό στην επόμενη συνάντησή μας στις 21 Ιουνίου. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε σταθεροποιήσει, θα έλεγα, με τον τρόπο με τον οποίο προτείνατε την κατάσταση. Α, κάποιος άλλος έχει ζητήσει το λόγο. Η κυρία Μουνίζ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμένα μου, μου φάνηκε κάπως ευνηδιαστικό αυτό το οποίο έγινε. Ορίστηκε ο εισηγητής, αποφασίστηκαν όλα αυτά τα είχαμε συζητήσει στους συντονιστές και άλλα είχαμε πει οι εκπρόσωποι, οι συντονιστέ των πολιτικών ομάδων. Ε, Κοιτάξτε τώρα να σα εξηγήσω. Ο κύριο Γκουαλτιέρη είναι από το δικό σα κόμμα και ήδη έχει διαπραγματευτεί αυτή τη συμφωνία. Αν υπάρχουν αντιρρήσει μπορούμε να επανέλθουμε στο ΣΕΜΑ, αλλά είχα την εντύπωση ότι η πρόταση είχε προέλθει και από εσά. Και γι' αυτό βιάστηκα να δώσω τον ρόλο του εισηγητή στον κύριο Μπρόκ για να μην καθυστερήσουμε άλλο. Δεν έχω αντιρρήσεις. Εγώ διαφωνώ για τη διαδικασία. Όταν από διαφορετικέ πολιτικέ πέργε συμφωνούμε όσον αφορά τον ορισμό ενό εισηγητού κλπ. κλπ ε, τι γίνεται. Έχουμε, τα βρήκατε εσεί λίγοι και ενώ έχουμε 7 πολιτικέ ομάδε. Εγώ ε, δεν είμαι επί τη αρχή ε, αντίθετο, αλλά θέλω να μάθω με ποια διαδικασία εσεί φτάσατε σε αυτήν την απόφαση. Είμαστε επιφορτισμένοι να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία αυτή και ο κύριος Μπρόκ και ο κύριος Γκουαλτιέρη, οπότε εγώ απλά επιβεβαίωσα τις εξελίξεις τις οποίες εμείς θεωρούμε ότι βρίσκονται στην τελική τους φάση. Κύριος Γκουαλτιέρη, θα μου επιτρέψτε μου να διευκρινίσω λίγο τη φάση στην οποία βρισκόμαστε. Στο διαβριμένο Προεδρείο της ΑΦΕΤ είχαμε ήδη επιφορτήσει τρία μέλη να διαπραγματευθούν με τα Εθνικά Κοινοβούλια για το θέμα αυτό εξ ονόματος της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Τώρα πλέον η πρόταση που γίνεται είναι να μετατρέψουμε σε ένα κείμενο πλέον τα αποτελέσματα αυτής της α, εμπειρίας και αυτό θα γίνει αντικείμενο συζήτηση την επόμενη εβδομάδα. Έχει περάσει ήδη από τους συντονιστές όλων των πολιτικών ομάδων η συζήτηση αυτή. Κοιτάξτε, ήμασταν ενήμεροι, ήμουν ενήμερος, αλλά θα ήθελα ακριβώς να ακούσουμε αυτά που είπατε, κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα, δημοσιονομικός κανονισμός εφαρμόσιμος στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγγήτρια η κυρία Μπρέντνερ το σχέδιο γνωμοδότησης απευθύνεται στην Επιτροπή Προϋπολογισμών η οποία θα πρέπει να το υιοθετήσει μέσα στον Ιούλιο. Είναι ένα θέμα που αφορά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεταρρύθμιση αυτή ακολουθεί την κανονική, την τακτική νομική διαδικασία στα πλαίσια δηλαδή της συναπόφασης και γι' αυτό απαιτεί αρκετό, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δίνω το λόγο στην κυρία Μπρέντνερ για την ομοθετική της πρόταση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι στους συντονιστές συζητήσαμε για το προηγούμενο θέμα προς υποστήριξη του κ. Μπροκ. Τώρα, όσον αφορά το κανονισμό, και θα μιλήσω στα αγγλικά, γιατί κάναμε όλο το κείμενο ε, στα αγγλικά. Ε, να με συγχωρέσετε λοιπόν που θα μιλήσω αγγλικά. Εν συντομία θα πω τις ιδέες που βρίσκονται από πίσω. Ε, οι σκιώδες συναντήθηκαν μαζί μου την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η συνάντηση. Ο βασικός στόχος είναι να αυξηθεί η ευελιξία και η ταχύτητα στην εκταμίευση της ε, βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπήρξαν κάποιες διατάξεις στο κείμενο, ιδιαίτερως για κατεπήγουσες ανάγκες και τη σχετική βοήθεια στην περίπτωση φυσικών καταστροφών κλπ. Αλλά θα θέλαμε να προσταθεί ότι ενδεχομένως θα μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις όπως αυτές στη Βόρεια Αφρική δηλαδή μετάβαση προς ένα δημοκρατικό καθεστώς, όπου εκεί θα θέλαμε να γίνει μια ταχύτερη αλλαγή ε, ε, στο επίπεδο της χρηματοδότησης. Ε, δεν πρόκειται για φυσικές καταστροφές, παρόλο που ορισμένοι συνέκριναν την κατάσταση αυτή με ένα πολιτικό τσουνάμι. Και συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να προσαρμοστεί ο κανονισμός για να μπορούμε να αντιδράσουμε και σε ένα πολιτικό τσουνάμι τώρα ο συντονισμός με τους διεθνείς δωρητές. Και αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί η Επιτροπή προτείνει να συσταθούν ευρωπαϊκά trust funds αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τη δυνατότητα να συστήσει τέτοια ταμεία. Και βεβαίως το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συστήσει τα δικά της Trust Funds. Πώς μπορούν να αντιδράσουν άλλοι δωρητές ή τα Ηνωμένα Έθνη και ποιος θα επιφοριστεί με τη διαχείριση αυτών των ταμείων. Ο εισηγητής ε, στην ομάδα προπολογισμού, η κυρία Γκρέσλε, είπε ότι μπορεί να επιφορτιστεί με αυτό μόνο η Επιτροπή και ενδεχομένω, ε, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ανοιχτοί και να πούμε ότι θα μπορεί να είναι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γιατί ορισμένε φορέ είναι δάνεια τα οποία δίδονται από αυτά τα trust funds ή σε ορισμένε χώρε ενδεχομένω. Ε, ε, άρα λοιπόν ε, δεν, θα είναι, δεν είναι μόνο η Επιτροπή, αλλά και χώρες μέλη ή ιδιωτικές τράπεζες μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα ευρωπαϊκά trust funds. Ε, γιατί στην περίπτωση αυτή υπάρχει μεγάλη εμπειρία, όπως είναι με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, πρόκειται λοιπόν για ένα νέο τομέα διεθνών σχέσεων και θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο εγγύς ε, μέλλον. Και επίσης υπάρχει το ζήτημα της μείωσης του διοικητικού άχθους, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τρίτες χώρες όταν δεν ε, ήταν σε θέση να εκπληρώσουν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το θέμα της διαχείρισης του κινδύνου. Εν συντομία θα διατρέξω ορισμένες τροπολογίες για να φωτίσω ορισμένες από αυτές και να σας εξηγήσω. Υπάρχει μια τροπολογία της κυρίας Γκρέσλε στη περίπτωση των ανθρωπιστικών κρίσεων και καταστροφών που συμβαίνουν μετά την 1η Δεκεμβρίου του έτους προπολογισμού. Ενδεχομένως εδώ η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια του επόμενου έτους τα κονδύλια λοιπόν του επόμενου έτους. Ε, δεν είμαι βέβαιη ότι αυτή είναι μια καλή ιδέα. Ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε γιατί κάτι τέτοιο θα επέτρεπε κατά την άποψή μου στην Επιτροπή να, όχι να πιέσει τις χώρες μέλη να δώσουν χρήματα, αλλά να πάρει τα χρήματα του επόμενου έτους. Και ξέρετε, το περιθώρια είναι πολύ στενά κάθε χρόνο. Ε, και σχεδόν ποτέ δεν είναι αρκετά τα χρήματα. Νομίζω ότι θα ήταν ένας εύκολος τρόπος για την Επιτροπή ε, να βρει μια λύση, αλλά θα μας οδηγούσε μια δυσχερή ε, κατάσταση. Άρα λοιπόν έχω κάποιες επιφυλάξεις, αλλά πραγματικά είμαι ανοιχτή και σε άλλες γνώμες, δεν ξέρω. Επίσης το θέμα για το ποιος έχει το δικαίωμα, ποιος έχει τις αρμοδιότητες εφαρμογής. Αυτή είναι μια συνέπεια τη ε, σύσταση τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, που είπαμε ότι είναι υπεύθυνη για το δικό τη ε, προπολογισμό. Αλλά ορισμένε φορέ στι αντιπροσωπείε ε, δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν υπάρχει επαρκές ε, προσωπικό και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ε, ρωτάει κατά πόσο θα έπρεπε να εκχωρήσει την αρμοδιότητα αυτή για πρακτικού λόγου στην Κομισιόν. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο αντίθετο επιχείρημα. Επίση, υπάρχει ένα άλλο θέμα τη ΑΦΕΤ, ένα παλιό σημείο, μία άδεια για μία γραμμή του προπολογισμού. Um, Επίση, το θέμα τη υποστήριξη του προπολογισμού. Η κυρία Γκρέσλε έχει υποβάλει εδώ αρκετά περιεκτικέ τροπολογίε. Υπάρχει μια πράσινη βίβλο αυτή τη στιγμή και η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει περιεκτικέ προτάσεις. Δηλαδή, εάν θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση με όλα αυτά τα λεπτομερικά τμήματα για την υποστήριξη του προπολογισμού ή να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδικά μια διαδικασία για την υποστήριξη του προϋπολογισμού και ίσως να περιμένουμε όλα αυτά πριν λάβουμε τη σχετική απόφαση. Δηλαδή ε, ε, ε, θα το παραλείψουμε ή όχι όσον αφορά την υποστήριξη του προϋπολογισμού ζητάει να ενισχυθούν τα εθνικά κοινοβούλια για να μπορούν να ασκούν τον έλεγχο και επίσης μη κυβερνητικοί οργανισμοί γιατί ε, σε πολλές χώρες όπου υπάρχει διαφθορά τα, και τα κοινοβούλια είναι διεφθαρμένα. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα κοινοβούλια αυτά που μπορούν να ενταχθούν στην ε, κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε σε αυτά. Επίσης υπάρχει ε, ε, μια κεντρική βάση δεδομένων που συστήνεται και που υπάρχουν ιδιώτες, ή οργανισμοί οι οποίοι έχουν αποτύχει στην ε, εφαρμογή, στην εξοποίηση των κονδυλίων και έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το μαύρο κατάλογο για να μην τους χορηγηθούν πλέον άλλα χρήματα. Ενδεχομένω είναι δύσκολα τα πράγματα για τις τρίτες χώρες εκεί που δεν υπάρχει καμία προστασία των δεδομένων αλλά θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι υπάρχει μια τροποποίηση ούτως ώστε να υπάρξει και σε αυτές τις χώρες, μια τροποποίηση για τις χώρες όπου υπάρχει κάποια προστασία δεδομένων. Και ένα άλλο σημείο στο οποίο αναφέρουμε στην αιτιολογική σκέψη για τις ε, δαπάνες ε, που είναι επιλέξιμες ε, ε, περιπτώσεις που μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι, δηλαδή καταπήγουσες ανθρωπιστικές ε, περιπτώσεις ε, και θα θέλαμε εδώ να προσθέσουμε μια κατάσταση η οποία συνιστά μια απειλή για τη δημοκρατία ή απειλή να κλιμακωθεί σε μια σύγκρουση. Πιστεύω θα πρέπει να γίνει εδώ αυτή η προσθήκη. Αυτά είναι κάποια σημεία τα οποία θα ήθελα εδώ να φωτίσω και αναμένω τα δικά σας σχόλια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκουαλτιέρη έχει στήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η πρόταση την οποία μας προτείνει η κυρία Μπρέντνερ είναι πάρα πολύ καλή έκθεση γιατί αντιμετωπίζει ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα το πρόβλημα του δημοσιονομικού κανονισμού. Προσπαθεί να συνδυάσει δύο αντιτιθέμενες, αντιφατικές μεταξύ τους, αν θέλετε, κατευθύνσεις. Από τη μία τον αναλυτικό έλεγχο των διαδικασιών που επιτρέπουν στην αρχή επί του προϋπολογισμού να επαληθεύει πάντα την σωστή και χρηστή χρήση των πόρων της Ένωσης και από την άλλη, και αυτή είναι και μια πάρα πολύ σημαντική απέτηση θα έλεγα, να διασφαλίσει την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα, επικαιρότητα και χρησιμότητα στην χρήση των πόρων. Και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρόταση της κυρίας Γκρέσλε, εισηγήτρια στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, προσφέρουν θα έλεγα διαφορετικές μορφές αντιμετώπισης, κάλυψης των αναγκών και οι δύο είναι θα έλεγα πιστικές αλλά παρόλα αυτά έχουν και κάποιες αδυναμίες. Γι' αυτό ακριβώς η πρόταση την οποία μας καταθέτει η Φρανσίσκα Μπρέντνερ προσπαθεί να καλύψει τις αδυναμίες των προηγούμενων εγγράφων με κάποιες προτάσεις τις οποίες γενικά θα έλεγα εμείς μπορούμε να δεχτούμε. Και η χρήση των μη χρησιμοποιημένων πόρων μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, τα λεγόμενα καταπιστεύματα, τα trust funds, βάζοντας κάποια όρια λιγότερο δεσμευτικά από αυτά τα οποία προτείνει η Γκρέσλε, αλλά εν πάση περιπτώσει και τη δυνατότητα πόρων από τον ιδιωτικό χώρο. Δυνατότητα εκ των προτέρων κάλυψης ορισμένων αναγκών στην περίπτωση κρίσεων, όχι μόνο ανθρωπιστικών κρίσεων, αλλά θεμάτων που έχουν σχέση και με πολιτικές κρίσεις, και όχι μόνο φυσικές καταστροφές και ταυτόχρονα τα θέματα των διαγωνισμών και του ρόλου των τρίτων χωρών προσπαθώντας να περιορίσουμε δηλαδή το συνολικότερο κόστος. Λοιπόν, συνολικά οι προτάσεις Μπρέντνερ είναι καλές. Ε, στηρίζω ιδιαίτερα και την τροπολογία που αφορά ένα επιπλέον βήμα γύρω από την διαφάνεια. Εμείς ε, έχουμε σαν στόχο να συμπληρώσουμε τις προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ένα άλλο θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι σχετικά προβληματικό και το οποίο δεν αναφέρεται στο κείμενο της κυρίας Μπρέντνερ είναι η τροπολογία την οποία κάνει η Γκρέσλε στο άρθρο 55 στον δημοσιονομικό κανονισμό. Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής του προϋπολογισμού από την Επιτροπή, από το προσωπικό της Επιτροπής υπό τον έλεγχο των αρχηγών προϋπολογισμών, των αρχηγών των αντιπροσωπιών, των υπευθύνων των αντιπροσωπιών. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ή έχουμε να κάνουμε με μια επιπλέον αρμοδιότητα των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Αντιπροσωπείας. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να το δεχτούμε. Αν από την άλλη θέλουμε να μειώσουμε τις αρμοδιότητες των αρχηγών αντιπροσωπιών, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 58, αν άκουσα καλά, στην ουσία έχουν ε, την δυνατότητα να ελέγξουν και όχι απλά να εκτελέσουν μία δαπάνη, τότε σε αυτή την περίπτωση τροποποιούμε επί της ουσίας την ευαίσθητη θα έλεγα ισορροπία στην οποία έχουμε καταλήξει στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Λοιπόν, δεν είναι πρόθεσή μας να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά ίσως θα πρέπει να αναδιατυπώσουμε κάπως τα πράγματα για να μην υπάρχουν παρανοήσεις και δυσκολίες κατανόησης γενικά. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιέρη. Νέμσκι. Σκιώδη εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γκρέσλε και την κυρία Μπράντνερ για την προσπάθειά τους σχετικά με τη σημασία καθορισμού των σωστών κανόνων για τη διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις προτάσεις του καθοδηγεί σωστά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διασφαλίζει τη σωστή, ε, θα έλεγα, χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Υποστηρίζω την πρόταση της κυρίας Μπραντνερ να υπάρξουν ξεχωριστές γραμμές για τον προϋπολογισμό για κάθε ε, αποστολή και πά, για κάθε δράση συγγνώμη και πά. Υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ μας για τον δημοσιονομικό κανονισμό. Νομίζω ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να διαχειριστεί τα μελλοντικά ευρωπαϊκά καταπιστεύματα. Κανένα άλλο σώμα δεν θα έχει έλεγχο σε αυτά τα καταπιστεύματα. Μόνο τότε θα, θα διασφαλιστεί η αποτελεσματική τους χρήση. Και θα πω στην κυρία Γκρέσλε ότι οι ιδιωτικές τράπεζες δεν μπορούν να λειτουργούν σαν διαχειριστές με εξουσιοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αναφερόμεθα στα χρήματα των φορολογουμένων μας. Θα είχα και άλλα σχόλια εδώ, αλλά θα ήθελα να μας πει η κυρία Μπραντνερ τι διευκρινήσεις μπορεί να μας δώσει στον τομέα αυτό. Σχετικά με την τροπολογία για το άρθρο 53 για τις εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή του προϋπολογισμού προς το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι πέρυσι καταλήξαμε σε μια συμφωνία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επιτρέπει την διαχείριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής να γίνεται από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, Λοιπόν, τώρα το να προτείνει κανείς μια διαφορετικού τρύπου επανεξουσιοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν κατάλαβα καλά, αν κατάλαβα καλά, αυτό μου θυμίζει και τις την τροπολογία 10 στο 120, υπό παράγραφος 2 και εκεί αναφέρεται σε αναδρομικές καλύψεις ποσών σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική προστασία και καταστάσεις οι οποίες απειλούν στο να κλιμακωθούν σε ένοπλες συγκρούσεις. Γιατί απαιτείται αυτή η απαρίθμηση εδώ. Ο όρος ένοπλη σύγκρουση περιλαμβάνεται ε, στον ορισμό κατεπήγουσα ανάγκη ή δεν υπάρχει μια τέτοια συμπερίληψη. Αναφέρομαι εδώ στην άμεση χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας για κάλυψη ανθρωπιστικών αναγκών στη Λιβύη και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, ακόμα και αν δεν υπήρχαν ε, λέξεις όπως ένοπλη σύγκρουση στο αρχικό νομοθετικό κείμενο με βάση το οποίο λήφθηκε η απόφαση. Ευχαριστώ κυρία Νέμσκι. Η κυρία Γέτεν Μάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Φραντσίσκα Μπραντνερ για την καλή, για το καλή της εργασία και την καλή συνεργασία. Η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας ήταν πραγματικά πολύ καλή και νομίζω ότι όλοι την χρειαζόμαστε. Και πιστεύω ότι αυτό δείχνει ότι η ΑΦΕΤ, η Επιτροπή μας, θα πρέπει εν γέννη να εστιάσει περισσότερο σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τον προϋπολογισμό, τον, την ε, εφαρμογή του, τη χρησιμοποίησή του ή ε, και άλλα θέματα που αφορούν τις ε, διαδικασίες του προϋπολογισμού. Εγώ υποστηρίζω την, τις προαθήσεις από την κυρία Μπραντνερ τροπολογίες αλλά θα ήθελα να πω ότι προσωπικά είμαι κάπως επιφυλακτική όσον αφορά την απευθείας υποστήριξη του προϋπολογισμού. Δεν είμαι βέβαιη κατά πόσο η έκθεση αυτή είναι δεδομένο τόπος να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι μελλοντικά θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα χρήματα πηγαίνουν ε, ε, εκεί που θα έπρεπε ακριβώς ε, να πάνε. Ενώ δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και αυτό αφορά ζητήματα εφαρμογή εκτέλεση του προπολογισμού. Επίσης θα ήθελα να απαντήσω το ζήτημα που έθεσε η κυρία Πράντνερ για τη χρησιμοποίηση χρημάτων από τον προπολογισμό του επόμενου έτους. Εγώ είμαι κάπως επιφυλακτική και θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο αυτό το θέμα γιατί φοβούμε ότι ενδεχομένως το Μάρτιο με τον τρόπο αυτό να αδειάσει ε, ο προπολογισμός, να μην υπάρχουν πια χρήματα. Τώρα, όσον αφορά κάποιες άλλες τοπολογίες που εγώ κατέθεσα για το άρθρο 31, παράγραφος 2, επί παραδείγματι, όπου θα ήθελα να προτείνω μια μεγαλύτερη διαφάνεια, ούτως ώστε να υπάρχει ε, ενημέρωση, να υπάρχει πληροφόρηση σχέση με τη χρησιμοποίηση των ε, κονδυλίων και επίσης σε σχέση με τα αποτελέσματα, γιατί νομίζω ότι οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τα αποτελέσματα και πώς χρησιμοποιούνται τελικά τα χρήματα αυτά. Και ε, με τον τρόπο αυτό και θα αντιφερθούν περισσότερο για ζητήματα της αναπτυξιακής βοήθειας. Τώρα, μια άλλη τροπολογία αφορά το άρθρο 88. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στο ζήτημα ε, κακής χρήσης του προϋπολογισμού, εκμετάλλευσης του προπολογισμού, Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο δίδεται ένα ορισμένο ποσό χρημάτων στην κυβέρνηση της Παλαιστίνης και τελικά ή στα μισά του χρόνου υπάρχει ένας καινούριος προϋπολογισμός. Και ξέρουμε ήδη στι αρχέ του χρόνου ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να συμβεί. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια μορφή εκμετάλλευση ή κακοδιοίκηση. Και ενδεχομένω υπάρχουν και άλλα θέματα. Που γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει στις αρχέ του χρόνου να προσπαθήσουμε να ξέρουμε πώ θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα γιατί βεβαίω ενδεχομένω μπορούν να κύψουν κάποια θέματα τα οποία δεν είμαστε θέσει να τα γνωρίσουμε εκ των προτέρων. Αλλά στην περίπτωση αυτή, για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο έχει επαναληφθεί για πολλά χρόνια και όλοι το γνωρίζουν. Παρόλα αυτά, ε, δεν γίνεται τίποτα. Ευχαριστούμε. Κυρία Μπραντνερ, θέλετε να κάνετε κάποια τελικά σχόλια. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια που πραγματικά ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα. Ε, θα πάρω με τη σειρά τις ερωτήσεις. Καταρχήν για τον κύριο Γκουαλτιέρη. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια σας και μοιράζομαι τις ανησυχίες για το άρθρο 55 που είναι αυτό που αφορά το προσωπικό της Επιτροπής και της και την ε, υποπτή εκ μέρους της επικεφαλής των αντιπροσωπιών. Ε, αν έχετε κάποια πρόταση θα σας ήμουν ε, ευγνώμων. Εάν ε, θέλετε να μου δώσετε ένα κείμενο, νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο. Γιατί πραγματικά συμμερίζομαι τι ανησυχίε ότι μπορεί ενδεχομένως να υπάρξει μια λαμφασμένη ερμηνεία εδώ. Κύριε κυρία νομίζω ότι όσον αφορά τα trust funds, τα καταπιστεύματα, Συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλε. Είμαι πολύ κατά της ε, χρήσης των ιδιωτικών, ε, της των ιδιωτικών τραπεζών, για παράδειγμα. Αλλά νομίζω ότι από την άλλη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να είναι ε, ένας παράγων, γιατί έχουν την εμπειρογνωμοσύνη, γιατί ξέρουν πώς πρέπει να το κάνουν ε, χωρίς να πάνε υπερβολικά μακριά. Επίσης αναφερθήκατε στο 53-4. Εδώ το θέμα είναι ότι η Επιτροπή έχει εκχωρήσει λειτουργικές ε, δαπάνες από τις επικεφαλής των αντιπροσωπιών στις υποεπιτροπές. Ε, ε και ο προβληματισμός καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αλλά το feedback από ορισμένε αντιπροσωπείε είναι ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό γιατί δεν έχουν αρκετό προσωπικό ε, στην υπηρεσία αυτή ε, και θέλουν να το εκχωρήσουν στην Επιτροπή. Ε, ε, αυτό είναι αστείο γιατί η Επιτροπή πάλεψε πραγματικά για να έχει αυτό το δικαίωμα και τελικά ε, διαπιστώνει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό στο επίπεδο πολλών χωρών. Και τελικά επαναχωρούν σε σχέση με αυτό το οποίο είχαν αποφασίσει αρχικά. Επίσης θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση για το 120 το κείμενο λέει καταστάσεις που απειλούν να κλιμακωθούν σε ένοπλες σειράξεις. Δηλαδή η βασική ιδέα είναι ότι δεν πρόκειται για ένοπλες σειράξεις, αλλά για απειλή, για, για καταστάσεις που, που, που ενδεχομένως θα κλιμακωθούν. Ε, ε, δηλαδή μια κρίση που βρίσκεται υπό εξέλιξη και όταν κλιμακωθεί μια κρίση η ιδέα είναι ότι είναι πολύ αργά για μια παρέμβαση. Ε, και τότε δεν είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε με ταχύτητα και με έναν ευέλικτο τρόπο. Η βασική ιδέα λοιπόν είναι να αντιδράσουμε στο επίπεδο της ε, πρόληψης όταν υπάρχουν ενδείξεις τα πράγματα πηγαίνουν προς την λάθος κατεύθυνση ούτως ώστε να μπορούμε να δράσουμε ε, ταχαίως και να αποφύγουμε να εμποδίσουμε την ένοπλη σύραξη. Αυτή είναι η βασική ιδέα της πρόληψης λοιπόν. Ελπίζω ότι είναι χρήσιμη αυτή η διευκρίνηση. Για τις δικές ανησυχίες συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να συζητάμε για τα, και σημαντικό συζητάμε για τα θέματα προπολογισμού. Και εγώ έχω το ίδιο θέμα για την υποστήριξη του προπολογισμού. Ε, νομίζω ότι είπατε ότι καλό είναι να το αφήσουμε απ' έξω και να υπάρξει μια διαδικασία στο επίπεδο της ε, ΔΕΒΕ με την Επιτροπή και τις χώρες μέλη και ίσως να μην προδικάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Ίσως μπορείτε να καταθέσετε μια τροπολογία διαγραφής αυτού του ε, ε, κειμένου. Εγώ συμφωνώ. Για το άρθρο 31, όσον αφορά τη διαφάνεια, προτείνω όχι μόνο οι καλυπτόμενοι, ευεργετούμενοι, αλλά όπω είναι τώρα για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ καλή για το άρθρο 38 όσον αφορά το τροποποιητικό, το τοπικό σχέδιο προπολογισμού. Εγώ ε, έχω διχαστεί για αυτές τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή καταγράφει αυτού, αυτού του τροποποιητικού σχεδίου προπολογισμού, παρά το ότι προβλέπεται και καταρχήν θεωρητικά όμω, κύριε Χέσλε που είναι η συγγεντρία, θέλει να έχει υπάρχει ένα και μόνο τροποποιητικό σχέδιο προπολογισμού. Όμω πάλι μου φαίνεται αυτό πάρα πολύ υπερβολικά στεγανό, γιατί ίσω σε κάποιε περιπτώσει κανεί χρειάζεται δύο διαφορετικά σχέδια προπολογισμού. Να βρούμε επομένω κατόπιν μετά ένα συμβασμό μεταξύ των δύο, και να υπάρχει κάποιο περιορισμό γιατί όπως τώρα το σύστημα δεν είναι στεγανό έναντι των καταχρηστικών ε, ε, ε, χρήσεων όπως είπε του προπολογισμού. Άρα θα πρέπει και εμείς να σταματήσουμε αυτή την καταχρηστική επίκληση του προπολογισμού αυτά για την πρότασή μου. Επίσης, η κυρία Κρέσλε, νομίζω ότι έδειξε πνεύμα συνεργασίας και θεωρώ ότι το κείμενο αυτό είναι μακροσκελέστατο και γι' αυτό έχουμε την άλλη μεριά λίγες τροπολογίες άρα επετέλεσε άριστο έργο τα πήγε πάρα πολύ καλά ε, οπότε λίγες μικρές μεταβολές μόνο υπάρχουν εντάξει δεν, δεν έχει διατελέσει για πολύ καιρό ε, μέλος της Επιτροπής ε, της Εξωτερικής Σχέσης πάντως συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά αγαστή συνεργασία και ελπίζω θα τα καταφέρουμε και επίσης συμπαθάτε με για την πίεση χρόνου αλλά ε, τι να κάνουμε. Πάντω τα πάμε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι θα βοηθήσουμε πάρα πολύ το έργο τη Επιτροπή των Προπολογισμών. Ευχαριστώ κυρία Μπράντνερ. Ο προπολογισμό προβλέπει την 17η Ιουνίου την παρουσίαση των τροπολομιών στις 12 και στις 21 Ιουνίου την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Περνάμε στο τελευταίο θέμα που προβλέπεται στη σημερινή μας συνεδρίαση, έκθεση Μπέλντερ για τις σχέσεις με το Ισραήλ σχετικά με την επίσκεψη την οποία έκανε ο κύριος Μπέλντερ 24 με 26 Μαΐου στο Ισραήλ. Δίνουμε την δυνατότητα, όπως ξέρετε, στους Προέδρους των διαφόρων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών να παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους για τις επισκέψεις τις οποίες έχουν κάνει. Πρόσφατα ακούσαμε και την έκθεση του κυρίου Ντερόσα για την επίσκεψη στην αντιπροσωπεία στη συνάντηση μάλλον με το νομοθετικό συμβούλιο της Παλαιστίνης και σήμερα έχουμε την ομόλογη θα έλεγα περίπτωση του κυρίου Μπέλντερ ο οποίος αυτός επισκέφτηκε τους αντίστοιχους θεσμούς του κράτους του Ισραήλ. Θα σας ακούσουμε με ενδιαφέρον. Έχετε το λόγο κύριε Μπέλντερ. Μπέλντερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. 23 με 26 Μαΐου του 2011. Ε, εργαστήκαμε στην αντιπροσωπεία μας για σχέση με το Ισραήλ. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Τα μέλη της αντιπροσωπείας μπόρεσαν να εξοικειωθούν με τα προβλήματα της ε, Ισραηλιτικής κοινωνίας. Πολύ ενδιαφέρουσα βέβαια ήταν συνεδρίαση με τα μέλη της Κνεσέτ. Τρίτη, 23 Μαΐου, έγινε αυτή η συνάντηση. Είχαμε επίσης και τον ε, πρέσβη, τον κύριο Στάνλι, που είναι αντιπρόσωπος του ΟΗΕ. Αυτός έκανε την εισήγηση. Επίσης ε, διαπιστώσαμε την σταθερότητα της υπό τον κύριο Νετανιάχου κυβερνήσεως. Στη συνεδρίαση αυτή, συνάντηση με την Κνέσετ, ε, συζητήσαμε τα εξή. Συζητήσαμε για τον εκδημοκρατισμό τη Μέση Ανατολής. Οι Ισραηλινοί είπαν ότι προβληματίζονται όσον αφορά τις εξελίξεις σε Αίγυπτο και Συρία τις γείτονες χώρες τους. Δεύτερον, είχαμε την Παλαιστινιακή πρόταση για τον Σεπτέμβριο στην σύλληψη του ΙΕΒ, ώστε να ανακηρύξουν το κράτος τους. Όσον αφορά την, ε, αντιπολίτευση, υπήρχαν ε, πολλοί βουλευτές της Καντιμά, οπότε και είπαν να μην νομιμοποιήσει, να μην αναγνωρίσει την Χαμάς το Κοινοβούλιο. Ανησυχούν οι Ισραηλοί για την συμφιλίωση Χαμάς και Αλφατάχ. Επίσης, μιλήσαμε για το Ιράν, για στρατηγικά ζητήματα, για το Ισλάμ στην Ευρώπη, αλλά επίσης εφήγει και η εμπορική συμφωνία της Άκρα. Ο πρόεδρος της μας μίλησε για λίγο και είπε ότι το Ισραήλ τίνει χειραφιλίας και συνεννόησης προς τις γείτονες χώρες θέλει ειρήνη με όλες τις γείτονες χώρες όμως θεωρεί ότι διακυβεύεται το θέμα της ασφαλείας της χώρας. Όποιος δεν αμφισβητεί το δικαίωμα ύπαρξης της χώρας μπορεί να αποτελέσει συνομιλητή του Ισραήλ. 25 Μαΐου τώρα. Επισκεφτήκαμε το κέντρο απορρόφησης μεταναστών στο Ισραήλ. Μιλήσαμε με νέους που εργάζονται εκεί. Είπαν ότι βοηθούν την εγκατάσταση των μεταναστών. Θέλουν να υπάρξει κάποιο είδους εγκατάσταση των μεταναστών εκεί και υπήρξαν επίσης και κάποιες συζητήσεις για το ποδόσφαιρο στα σχολεία. να ε, είχαμε κάποιους περιήγες που θαυμάσαμε διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Είδαμε τι γίνεται εκεί με κάποιου είδου ε, περιπτώσεις παιδιών ε, του Ντονάσιλο και άλλων ε, μη προνομιούχων το ΣΥΠΗΝ οι οποίοι σπουδάζουν εκεί. Είχαμε επίσης και συνάντηση και με παιδιά που έχουν πέσει θύμα κακοποίησης. Η επιτυχία μας, η αποστολή αυτή στο Ισραήλ, θεωρώ ότι πέτυχε και ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους. Νομίζω ότι όλοι βοήθησαν. Η κυρία Πέρεθ επίσης βοήθησε, η Κριστίν Γκαρίγκ και ο Λάρς επίσης, Λάρς Βεβαίως και βοήθησαν όπως πάντα οι διερμηνείς μας. Ό,τι τυχόν ερωτήσει έχετε να τις απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει ο ομόλογος του κυρίου Μπέλντερ, ο κύριος Ντερόσα, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο. Κύριε Ντερόσα. Σας ευχαριστώ, κύριε Αλμπερτίνη. Ευχαριστώ και τον Μπαστιάν για την έκθεσή του όσον αφορά αυτή την επίσκεψη στη χώρα. Στο Ισραήλ είναι πολύ σημαντικό η ΑΦΕΤ να προχωρήσει σε εξέταση αυτών των εκθέσεων και εγώ σύνταξα μια τέτοια έκθεση όσον αφορά την ε, επίσκεψη της αντιπροσωπείας για την Παλαιστίνη. Να μην ξεχνούμε ότι ο πρόεδρος Μπούζεκ σήμερα βρίσκεται στο Ισραήλ. Επίσκεψη τετραήμερη έκανε και επίσης σήμερα επέπρωτο να συναντηθεί με μέλη της ε, Κνεσέτ διαμορφωθεί με μια ισορροπημένη ολοκληρωμένη γνώμη για το τι θα γίνει όσον αφορά με το Μεσανατολικό, πώς θα σταματήσει εκεί η κρίση. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο Πρόεδρος και επίσης επανέλαβε ότι χρειάζεται να γίνουν άμεσες επαφές μεταξύ Παλαιστινίων και των Ισραηλιτών, ούτω ώστε να φτάσουμε σε ειρήνευση και για να υπάρξει ειρήνευση στην περιοχή αυτή την ευρύτερη θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία Ισραηλιτών Παλαιστινίων για μια λύση που να εγγυάται δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, ακυριότητα του κράτους ε, και για τους μεν και για τους δε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά μην τα ξεχνάμε, τα τα έχουμε πολιτική συζήτηση σχετικά με το πρόβλημα και εγώ πιστεύω ακράδοντα ότι οι σημερινές προσπάθειες που καταβάλλονται από την σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ ώστε να ματιώσουν τη, τα διαβήματα του, του, της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ και την αγνώρισή τους προσπάθεια αυτή η Ισραηλινή νομίζω ότι είναι λάθος νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που πάνε να κάνουν οι Παλαιστίνοι να πείσουν ε, όποιον μπορεί να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις ευθύς αμέσως ο χρόνος πιέζει ο Μπαστιάν πήγε εκεί στην περιοχή και εγώ ο πρόεδρος του κοινοβουλίου μας και όλοι εμείς ε, το διαπιστώσαμε αυτό ότι ο χρόνος πιέζει. Ακόμα και αν καταφέρει το Ισραήλ να μπλοκάρει αυτή την ε, ε, προσωρινή μονομερή ανακήρυξη αυτό πώς θα ωφελεί στο Ισραήλ, πώς θα αγγίθει η ακυρότητα στο Ισραήλ, πώς θα φέρει την ειρήνη πιο κοντά. Άρα θέλω να πω όλοι εμεί να πείσουμε και τους μεν και τους δε να σοβαρευτούν, να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να επιλύσουν ό,τι θέματα ακόμα εγκρεμούν. Η Ένωση προτίθεται να βοηθήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν πρόκειται καμία εξίσωση. δεν, δεν, λέει πουθενά, δεν πουθενά γραμμένο ότι το προστασία των δικαιωμάτων των μεν συρρυκνώνται τα δικαιώματα των δε. Όμως είναι σίγουρο ότι χρειάζεται ειρήνη, χρειάζεται δημοκρατία, και αυτό είναι κάτι το χρειάζονται όλοι. Και η Ευρώπη το χρειάζεται και το Ισραήλ το χρειάζεται. Θέλουμε ως γείτονα του Ισραήλ δημοκρατική Παλαιστίνη. Αυτό θα είναι καλύτερη εγγύηση για την κυριότητα του κράτους και την ασφάλεια του του. Ευχαριστούμε κύριε Ντέρο, πρόεδρος. Ο ρόλος του έχει ο κύριος Βίγκενιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω... Σύντομη ερώτηση για τον κύριο Μπέλντερ. και για τη δυνατότητα συνέχισης των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ε, πλευρές οι οποίες δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το θέμα με μια κάποια ευολιξία. Ξέρουμε ότι πρόκειται για το Χαμάς. Θα ήταν δυνατόν από πλευράς του Ισραήλ να διαφοροποιήσει από τη μία τον Χαμάς και από την άλλη μια κυβέρνηση η οποία βέβαια έχει μέσα της και τη συμμετοχή του Χαμάς. Αυτό μπορεί να υπάρξει σαν λογική αρκεί μια κάποια ευελιξία από πλευράς του Ισραήλ. Ευχαριστώ κύριε Βίγκενινγκ. Ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την έκθεση που μας ανέλησε από την επίσκεψη ε, στο Ισραήλ. Περίμενα όμως, δεν ξέρω αν είναι ο χρόνος, είδα και τα γραπτά, κάποια αξιολόγηση μπροστά στο κρίσιμο θέμα που έχουμε σε σχέση με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Ακούστηκε στην έκθεση του συναδέλφου ως μια πρόταση των Παλαιστινίων. Δεν υπάρχει ένα αίτημα, δεν υπάρχει μια διεκδίκηση. Τι θα γίνει με τη Γενική Συνέλευση που, έχουμε, που έχει στο το ΟΗΕ το Σεπτέμβρη. Υπάρχει αντίδραση του ο, Ισραήλ. Θα τον παρακαλούσα αν μπορούσε να μας πει ποια είναι η εντύπωσή του, ποια θα είναι η αντίδραση τη Ισραηλινής κυβέρνηση Και δεύτερο, ε, προβλέπεται επίσκεψη για άλλη μια φορά προσπάθεια από το στόλο ελευθερίας επίσκεψη και σπάσιμο του αποκλεισμού της Γάζας. Πέρσι είχαμε ε, δραματικές εξελίξεις. Ποιες είναι φέτο οι προθέσεις της, Ελλην... της Ισραηλινής Θα έχουμε επανάληψη τη ίδια οξύτητα. Ε, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένο. Τον ευχαριστώ τον συνάδελφο αλλά σε κάποια θέματα θα ήθελα και τη εκτίμηση απεκόμισαν και μια αξιολόγηση των γεγονότων και πού βρισκόμαστε για τη λύση του Μεσοανατολικού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Χούντι. Στο πρόεδρε. Στη, στη Ραμάλα, στη Παλαιστίνη ε, πήγαμε και, και, και στο κράτος και ήρθα αφού με εντυπωσίασε το τι, τι, τι ισχύει τον κόσμο στην ε, Παλαιστίνη. Ε, αδιαφορία, καμιά ανταπόκριση δεν υπάρχει στις προσπάθειες που γίνονται. Τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που γίνονται προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ τίποτα. Ε, τίποτα δεν γίνεται όσον αφορά αυτή την Αραβική Άνοιξη, τι γίνεται στην Αίγυπτο, τι γίνεται όσον αφορά την ιδέα συμφιλίωσης. Το Ισραήλ είναι αρνητικό. Δεν δέχονται αυτές τις προτάσεις, αυτή την προστασία της συμφιλίωσης. Μια αρνητική στάση επίσης και όσον αφορά την πρωτοβουλία στον ΟΗΕ. Τους λένε ότι είναι ενέργεια μονομερής. Δεν είναι, είναι πολυμερείς. Πάνε στον ΟΗΕ για να διευθετήσουν μια διεθνή σύγκρουση. Έχουμε πει σε αυτή την κοινή διακήρυξη της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου με το Ισραήλ όσον αφορά ε, το ότι ασπαστήκαμε τις ελληνικέ θέσεις χωρίς καμία διαφοροποίηση έχουμε αυτή επομένω. Ε, έχουμε εδώ πέρα αυτά τα οποία στα συμφωνούμε ενώ αναλυτές ε, Ειρηνοποιεί διάφοροι, το, το κέντρο Τρούμα, το κέντρο Κάρτερ, όλοι αυτοί έχουν μιλήσει υπέρ αυτής της πρότασης συμφιλίωσης για, για Χαμάς και Αλφατάχ. Θεωρείται ότι έτσι θα εκδημοκρατιστεί η Παλαιστίνη, έτσι μπορεί να διενεργηθούν το 2010 εκλογέ και έτσι υπάρχει ανταπόκριση στη θέση του Ισραήλ και πρέπει να έχουν συνομιλητή για να μιλήσουν για ειρήνη. Τώρα έχουν, θα έχουν κάποιον, θα αποκτήσουν κάποιον συνομιλητή που να εκπροσωπεί όλο τον το λαό της Παλαιστίνης. Είναι επίσης επικίνδυνο το ότι τμήμα του Κοινοβουλίου λαμβάνει υιοθετεί τόσο ριζοπαστικές θέσεις, τόσο πολύ μεροληπτή, χωρίς καμία διαφοροποίηση υπέρ της μιας πλευράς. Τι γίνεται με αυτές τις άμεσες ε, που πρότειναν οι Παλαιστίνοι πέρσι και ζήτησαν μόνο απλώς να υπάρχει κάποιο πάγωμα Στου στους, ε, στους εγκαταστάσεις, καταβλισμούς, στους Και για τη Χαμάς είπαν όχι. είπαν ότι είναι μονομερής η κίνηση το διάβημα στο νοιε Δεν έχουν αφήσει καμιά διέξοδο. Τίποτα δεν κάνουν για να ανταποκριθούν στην διεθνή δυναμική. έχουν φέρει εμπλοκή εδώ και χρόνια. Μονομερός μιλάνε για τα σύνορα του 67 και χειρότερα αφού συνεχίζουν για την οικοδόμηση του τείχους. Τι έγινε με τη συμφωνία της Γενέβης του 49 συνέχεια την παραβιάζουν οι Ισραηλοί. Ευχαριστώ κύριε, Πρόεδρε. Ε, δύο παρατηρήσεις. Εγώ θα σταθώ στο κοινό ανακοινοθέν που ε, υπάρχει μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας ε, του Κοινοβουλίου μας και τις συνομιλίες που είχαν με το Κοινοβούλιο, με την Κνεσέτ στο Ισραήλ και να εκφράσω και εγώ την ε, δυσαρέσκειά μου για το γεγονός ότι στο κοινό ανακοινωθέν εκφράζεται η άποψη ότι ε, η αναγνώριση του, του κράτους του, της Παλαιστίνης θα είναι μια... Ε, τέλος πάντων εκφράζεται η αντίθεση του Ευρωκοινοβουλίου στην αναγνώριση του κράτους της ε, Παλαιστίνης. Και εδώ δεν είναι ένα θέμα μιας μονομερούς ε, ενέργειας, όπως υπόθηκε και από τους ομιλητές πριν. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και από ό,τι έχω υπόψη μου δεν υπάρχει τέτοια τοποθέτηση του Ευρωκοινοβουλίου που να είναι αντίθετο σε μια τέτοια διαδικασία. Ω εκ τούτου δεν ξέρω ε, αν υπάρχει βάση για τους συναδέλφους να έχουν μια τέτοια ε, τοποθέτηση. Επίσης, θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στις τοποθετήσεις του Ευρωκοινοβουλίου ούτε στην πρακτική που υπήρχε μέχρι τώρα, η πρώτη τελευταία παράγραφο στο κοινό ανακοινωθέν, που, η οποία λέει ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή και το Ευρωκοινοβούλιο, δεν θα αποδεχτεί μια διαδικασία reconciliation ε, των Παλαιστινίων. Τέτοια γενική διατύπωση και ένα τέτοιος ε, τρόπος ε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, δεν είναι ισορροπημένο, δεν βοηθάει ε, την υπόθεση. Και τέλος, ε, οι αναφορές οι οποίες γίνονται στις ε, εξεγέρσεις στις ε, αραβικές χώρες και ο κίνδυνος για έναν ακραίο Ισλαμισμό ο οποίος θα μπορέσει να υπονομεύσει τις βασικές, τους βασικούς στόχους αυτών των εξεγέρσεων και αυτό το θεωρώ μια ε, παρέμβαση στα εσωτερικά ε, των χωρών αυτών και στις εξεγέρσεις που γίνονται ε, πολύ περισσότερο τέτοιοι κίνδυνοι προφανώς υπάρχουν δεν χωράει καμία αμφιβολία για αυτό το ζήτημα όμως πιστεύω ότι οι λαοί και οι δημοκρατικές δυνάμεις στις χώρες αυτές είναι αρκετά όριμες να ξέρουν οι ίδιες ποιους πρέπει να αφήσουν και με ποιους πρέπει να συμμαχίσουν σε μια διαδικασία ριζοσπαστικών αλλαγών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Eh, λοιπόν, ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλντερ, έχετε το λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση. Eh, eh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρατηρήσεις σας και τα σχόλια. Θα ήθελα να πω ότι μια αντιπροσωπεία έχει το δικαίωμα να εκφράσει τη δική της ε, θέση. Ε, αυτό συνέβη εδώ και δεν νομίζω ότι τους κανόνες ε, παραβιάστηκαν εδώ. Θεωρώ ότι εκφράστηκαν κάπως περίεργες απόψεις. Στο ένα κοινοβούλιο μπορούν να υπάρχουν, να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις. Τώρα όσον αφορά την σχέση μεταξύ Φατάχ και Χαμάσα. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Υπάρχουν βασικές αρχές του κουαρτέτου τις οποίες πάντοτε υποστηρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ καλείται η Χαμάς να είναι επικοδομητική και να προβεί σε διαπραγματεύσεις. Αλλά εξ όσων ε, γνωρίζω η Χαμάς εμένει στη θέση της της μη αναγνώρισης του κράτους του Ισραήλ και ε, συνεπώς ε, δεν θα υπάρξει καμία κίνηση. Όταν ε, μιλούμε για την, ε, την Αραβική Άνοιξη ε, και βλέπουμε τι γίνεται στην Αίγυπτο, θεωρώ ότι εκεί είναι μάλλον χειμώνα και όχι Άνοιξη. Εγώ ήμουν με μια αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο και πραγματικά κράτησα πολύ καλά ανοιχτά τα μάτια μου και τα αυτιά μου και θεωρώ ότι μπορούμε να μοιραστούμε τις ανησυχίες των Ισραηλινών σε αυτή την περίπτωση. Και θα ήθελα να τονίσω και πάλι, η αντιπροσωπεία μας ε, συναντήθηκε με εκπροσώπους της Κνεσέτ, οι οποίοι λένε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει μεταξύ Χαμάς ε, και Φατάχα είναι απαράδεκτο για αυτούς. Ε, μία συμφιλίωση δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει όσο η Χαμάς δεν κινείται η αναγνώριση του Ισραηλού κράτους θα πρέπει να γίνει. Ε, αλλιώς υπάρχει ένα διέξοδο και νομίζω ότι το Ισραήλ θα πρέπει να το επισημάνει και ε, πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα είπαν ότι ναι μεν επιζητούν την ειρήνη αλλά δεν είναι δυνατόν να κινηθούν με κλειστά τα μάτια. Ευχαριστώ κύριε Μπέλτερ Κλείνουμε τις εργασίες μας για σήμερα. Αύριο στις 9 έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικό της Ουγγαρίας. Ευχαριστώ.